Buenas Καλησπέρα σας. Σα καλησπέριζω όλε και όλους. Καταρχά να σα ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Να ευχαριστήσω όλους όσοι θα συμμετέχουν σε αυτή την ακρόαση που διοργανώνει η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών από την ε, Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των Ανθρώπου, από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική και ενδιαφέρουσα στιγμή για την πρωτοβουλία αυτή και βεβαίως επειδή έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ε, τους ομιλητές μας και τις ε, συζητήσεις ε, που θα γίνουν αργότερα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να μας χρησιμεύσει αυτό για τις καθημερινές μας εργασίες και τις εργασίες των διαφόρων υπηρεσιών στις διάφορες επιτροπές. Είναι η 15η επέτειος από την έγκριση του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για τις ε, γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια το ψήφισμα 1325 και θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν σημαντικό να εορτάσουμε αυτή τη στιγμή. Ε, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα 31 ε, Οκτωβρίου του 2000 για το ψήφισμα αυτό και ήταν ένα σημαντικό ε, σημείο καμπής για την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών σε ένοπλες σειράξεις και το πόσο δυσανάλογη είναι η κατάσταση αυτή για αυτέ. Στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μνήμα στα θέματα φύλου, στα θέματα που σχετίζονται με τις γυναίκες και το ψήφισμα αυτό καλύπτει σημαντικές πτυχές ε, ζητώντα μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, ε, μέτρα για την καταπολέμηση της βία λόγω ε, κατά των βιασμών και οποιασδήποτε άλλες μορφέ. Και πρέπει να σας πω ότι 15 χρόνια μετά ακόμα είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε τα ζητήματα αυτά, διότι ε, διαπιστώνεται ότι σε πολλές γωνιές του κόσμου εξακολουθούν ε, να υπάρχουν ε, ενεξελίξεις σειράξει και ζούμε φρικαλαιότητες και βιαιότητες και μεταχείριση και κακομεταχείριση ενώπιον των γυναικών και των νέων κοριτσιών. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό στο ψήφισμα αυτό είναι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ε, ανοικοδόμηση μετά το πέρας της σύραξης. Οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν ε, στην ε, επίλυση αυτών των σειράξεων και θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνέχεια στην εξέλιξη όλων των πολιτικών που σχετίζονται με την ανοικοδόμηση και στην επιστροφή της αξιοπρέπειας ε, για όλους τους πολίτες και κυρίως ε, για τις γυναίκες. Σε αυτή λοιπόν τη 15η επέτειο του ψηφίσματος ε, τα Ηνωμένα Έθνη καταρτίζουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του κειμένου και θεωρώ ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και να δούμε και τι μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να υπάρξει κατάλληλη εφαρμογή και αναθεώρηση του ψηφίσματος ε, και δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ψήφισμα. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στην φίλη και συνάδελφο Έλενα Βαλενθιάνο, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ Ράτσε που ε, μας προσκάλεσες ε, εδώ, να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ε, συζήτηση που θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι έχουμε μεταξύ μας ανθρώπους που δίνουν μάχη όλη τους τη ζωή ώστε να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος που πρέπει να διαδραματίζουν οι γυναίκες ε, για την επίλυση των σειράξεων και το πόσο υποφέρουν οι γυναίκες ε, στη διάρκεια της ιστορίας λόγω των πολέμων. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δύο ε, πτυχές. Είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα, αν και δεν είναι πολύ σωστό αυτό, και είμαστε και τα θύματα που πρωταγωνιστούν λιγότερο. Και αυτό είναι ένα χάσμα και πρέπει κάπως να το ε, διορθώσουμε το σφάλμα αυτό. Είναι όντως λοιπόν αυτή η 15η επέτειος του ψηφίσματος 1325 και έχει εγκριθεί ένα νέο κείμενο ε, για το μέλλον και η άποψή μου για την ε, εξέλιξη του ψηφίσματος ε, είναι αρκετά απεσιόδοξη. Θεωρώ ότι ελάχιστα καταφέραμε και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος βρίθει σειράξεων και οι γυναίκες είναι περισσότερο θύματα από ό,τι ποτέ και λιγότερο πρωταγωνίστρες από ό,τι ποτέ όσα ε, υπήρξαν από πλευράς νομοθεσίας ε, είναι ανεπαρκή, δεν μπόρεσαν να προστατέσουν τις γυναίκες και δεν μπόρεσαν να ε, βελτιώσουν τη συμμετοχή των, των γυναικών στη διάρκεια της ανοικοδόμησης. όλα όσα συμβαίνουν ανά τον κόσμο και θα μας πούν και οι προσκεκλημένοι μας αργότερα, είναι ότι το γεγονός ότι ορισμένες φορές όταν υπήρξαν γυναίκες οι οποίες βοήθησαν στον περιγυρό τους για να υπάρξει βελτίωση και ανοικοδόμηση μετά από το πέρας μιας σύραξης και ενός πολέμου, ε, είχαμε πάντα θετικά αποτελέσματα. Οι γυναίκες ε, στη διάρκεια της ιστορίας ήταν αυτές οι οποίες έπρεπε να φροντίζουν τους άλλους, ε, να τους προσέχουν, να τους θεραπεύουν και τίνουμε να έχουμε μία οπτική για τις ανάγκες των υπολείπων ε, που είναι αρκετά αληθινή και ξέρουμε ότι το να συμμετέχουν οι γυναίκες και για την επίλυση των ένοπλων σειράξεων και για τα συνδυνευτικές συζητήσει και ε, για την ανοικοδόμηση μετά από το πέρας των σειράξεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και παρόλα αυτά πολύ δύσκολα συμβαίνει. Επιπλέον και όταν εμφανίζονται και ριζοσπαστικά, ακραία και δολοφονικά φαινόμενα τον κόσμο, το φαινόμενο και παράδειγμα του Ισλαμικού κράτους και όχι μόνον αυτό, γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενο, είναι στόχος αυτός των ομάδων και των κινημάτων που είναι και σχεδόν στρατή του τρόμου. Οι γυναίκες και τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, κορίτσια είναι κατά προτεραιότητα στόχος ε, του Ισλαμικού κράτους, του Μπόκο Χαράμ και ξέρουμε ότι πρωτίστως είναι κατά των γυναικών και των παιδιών. Πρώτα αυτούς χτυπούν αυτές οι ομάδες. Και οι γυναίκες κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν ένα μέσο για να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή στην κοινωνία και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό μέσο, διότι ε, όταν... Ε, ελέγχου τις γυναίκες καταφέρνουν να ελέγχουν καλύτερα τον τοπικό πληθυσμό. Γι' αυτό και ακριβώς αποτελούν στόχο οι γυναίκες όλων αυτών των ακραίων και τρομοκρατικών ομάδων. Αυξήθηκαν λοιπόν οι πιέσεις προς τις γυναίκες, αυξήθηκαν οι κίνδυνοι για τις γυναίκες, αυξήθηκαν και τα θύματα φυσικά και γι' αυτό ακριβώς ε, ήγηκε η ώρα να εγκριθεί ένα νέο κείμενο από πλευρά Ηνωμένων Εθνών ώστε να δοθεί μια νέα όθηση στο ψήφισμα 1325, το οποίο κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια σημαντικά ε, στοιχεία και κάποιες σημαντικές εξελίξεις και ακόμα και μέσα στο ΝΑΤΟ έγινε μια απόπειρα να ανοιχτεί ένας χώρος για τις γυναίκες, ε, σαφώς όλα αυτά δεν αρκούν. Ε, ο ρόλος μας λοιπόν εδώ είναι να δώσουμε μια όθηση για τη συζήτηση, να συνειδητοποιήσει αφενός η κοινωνία τι συμβαίνει, αλλά και η κατάλληλη νομοθεσία είναι η άλλη πτυχή, και ε, τον, η εφαρμογή της νομοθεσίας στη συνέχεια είναι το τρίτο στοιχείο που είναι και το πιο δύσκολο ακόμα. Ε, στο Κοινοβούλιο βέβαια αυτό υπάρχει πολυφωνία, υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τελείως διαφορετικές ευαισθησίες, αλλά σήμερα θα θέλαμε με την ε, πρόεδρο της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ επίση, να δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένες να δώσουμε μια νέα όθηση στη συζήτηση ώστε να πάψουν καταρχάς να είναι οι γυναίκες θύματα και να αρχίσουν να είναι οι πρωταγωνίστριες. Να σταματήσουν λοιπόν πρώτα να είναι τα θύματα και ταυτόχρονα να γίνουν πρωταγωνίστρες στην ειρήνη. Να πάψουν να είναι θύματα του πολέμου και να γίνουν πρωταγωνίστρες τη ειρήνη. Αυτή είναι η πρόθεσή μα με την ακρόαση αυτή. Να σας καλεσορίσω όλους και να δώσω το λόγο και στην πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλεια και Άμυνα, την κυρία Φωτίγα. Uh, Κυρίε Πρόεδροι, κύριε και κύριοι, είναι για μένα μεγάλη τιμή να παρευρίσκομαι εδώ στην δημόσια ακρόαση για το ζήτημα της κατάστασης των γυναικών στις εμπόλεμες ε, περιοχές. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας. Επομένως, η κύρια μας, το κύριο αντικείμενο της Επιτροπής μας είναι οι ένοπλες συγκρούσει, καθώς επίσης και ε, τα προβλήματα των γυναικών στο πλαίσιο αυτών συγκρούσεων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 1325 το 2000 μετά από φρικτά εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια των πολέμων στα Βαλκάνια. Θυμόμαστε όλοι την Σρεμπρένιτσα ή τη σύγκρουση στη Ρουάντα και άλλες συγκρούσεις. Τότε λοιπόν, μετά από αυτά τα γεγονότα, είχαν εγκριθεί ε, μια σειρά από πολιτικά έγγραφα για τα ζητήματα αυτά. Και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κατά των κοριτσιών, και την ε, σχέση της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και της καταπολέμησης της βίας στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και στο πλαίσιο του διεθνού ε, ποινικού δικαίου, θα επίσης και του διεθνού ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σχετικά ψηφίσματα έχει θετήσει και η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κατάγομαι από την Πολωνία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα και ζω ακόμα στην Πολωνία. Γεννήθηκα επί του κομμουνιστικού καθεστώτος και είχα ίδια εμπειρία των παραβιάσεων των δικαιωμάτων που διαπράττονταν τότε υπό το ε, κομμουνιστικό καθεστώς. Με τα ίδια μου τα μάτια το είδα και ακόμα περισσότερο επειδή είμαι καθολική. Και αντιλαμβάνομαι και προσωπικά τα ζητήματα αυτά, τα παρακολουθώ. Παρακολουθώ τη στάση του Βατικανού στα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι το Βατικανό έχει αναγνωρίσει και έχει καλωσορίσει το ψήφισμα 1325. Ο Τελικός Νούντσιος πρόσφατα ε, ε, εξέφρασε τις απόψεις του επί τα θεμάτων αυτών. Το ψήφισμα 1325 καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων. Και αναφέρει ότι οι γυναίκες είναι εκείνε που υφίστανται τις μεγαλύτερες επιπτώσεις ε, στη ζωή τους από μια ενόπλη σύγκρουση. Οι γυναίκες και τα κορίτσια, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα ενός πολέμου, θύμα ενός πολέμου. Το ψήφισμα 1325 επίσης αναφέρεται στη σημασία που έχει ο ρόλος των γυναικών να ενισχυθεί στον τομέα της διατήρησης της ειρήνης, των ερευνευτικών αποστολών, καθώς επίσης και της ανοικοδόμησης μετά από έναν πόλεμο. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τομεί και κατά τη διάρκεια ενός μεγάλη χρονική περίοδου που οι γυναίκες μπορούν να συνεισφέρουν σε μια. Ε, ξεπέρασμα πολεμική σύγκρουσης. Χαίρομαι γιατί όλοι οι ομιλητές που έχουμε καλέσει σήμερα εδώ είναι ιδιαίτερα ε, καλοί γνώστες των θεμάτων τους, ιδιαίτερα των ζητημάτων ε, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, των ζητημάτων των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ταγματάρχη Στέφαν Καμιλέρη, για το πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Και στο δεύτερο μέρος της συζήτησή μας θα ακούσουμε από αξιωματικό του ε, στρατού της Μάλτας που έχει ε, μεγάλη εμπειρία έχοντας υπηρετήσει σε δύσκολες περιοχές, στο κέρας της Αφρικής, στα Βαλκάνια, στο επιχειρησιακό κέντρο ε, στην Αταλάντα, σε και στα κέντρα επιχειρησιακού σχεδιασμού στο Ηνωμένο στη Μάλτα και αλλού, τα οποία σχεδιάζουν ε, ειρηνευτικέ αποστολέ. Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνο επιχειρησιακού σχεδιασμού για το, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με χαρά θα ακούσω λοιπόν την παρουσίαση του Ταγματάρχη Καμιλέρη. Bueno, pues vamos Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παρουσιάσεις ε, των επιρογνωμόνων ε, στο πρώτο πάνελ. Ε, ήδη σας έχουμε ευχαριστήσει για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Γνωρίζετε ότι έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά για την αρχική σας παρέμβαση και όταν θα ακούσουμε τις πρώτες τρεις παρεμβάσεις, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές και στη συνέχεια, ε, εάν μας ε, φτάνει ο χρόνος, θα μπορέσουν να απαντήσουν οι ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Σάρα Λίνβαλ, που είναι ε, εκπρόσωπος ε, του Ιδρύματος Συρία Κβίνα. η έδρα τους είναι στο Λίβανο, αλλά είναι υπεύθυνη για τη Συρία. Η κυρία Λίνβαλ μπορεί να σας μιλήσει για την εμπειρία της την ε, οργάνωση γυναικών ε, ε, στην οποία εργάζεται και για το τι ακριβώς κάνει στη Συρία η οργάνωση αυτή. Συμμετείχε και στις συζητήσεις της προηγούμενης εβδομάδας στα Ηνωμένα Έθνη για την αναθεώρηση του ψηφίσματος 1325 και είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσει να μας διαβιβάσει ε, μέσω της εμπειρίας και των γνώσεών της ε, μια εικόνα της πραγματικότητας που ζουν ε, χιλιάδες γυναίκες σήμερα στην Συρία. Μια χώρα που αποτελεί παράδειγμα της φρικαλαιότητας και της βιαιότητας και των απάνθρωπων συνθηκών όπου ζουν πολλές γυναίκες. Κυρία Λίνβαλ, έχετε το λόγο. Thank you. Um, Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ε, σε ένα σημείο θα ήθελα να εστιάσω σήμερα, σε ό,τι αφορά την ανάληψη ενό ενεργού ρόλου από την πλευρά των ε, γυναικών. Θα αναφερθώ στο παράδειγμα της ε, Συρίας, αλλά βέβαια ε, δεν θα περιορίζομαι μόνο στο, στη Συρία. Θεωρώ πως το ψήφισμα 1325 είναι πραγματικά ένα ορόσημο σε ό,τι αφορά τον ενεργό ρόλο των ε, γυναικών. Ε, ε, και σε ό,τι αφορά την έμφαση που δίνουμε στην σεξουαλική διασφάλιση των γυναικών, νομίζω πως τώρα έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε το πόσο εκτεταμένη είναι. Τώρα αρχίζει να ανακύπτει γιατί και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται περισσότερο τι συμβαίνει. Η τελευταία έκθεση σε ό,τι αφορά τα στρατόπεδα βιασμών στον ε, Νότιο ε, Σουδάν, ειδικότερα αφού είχαμε ε, και μια διεθνή παρουσία που είχε ιδιαίτερη εντολή να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό. Δεν ξέρω αν έχει δει κανένα την ε, ταινία του 1982 του Κόνα του Βάρβαρο. Εν πάση περιπτώσει ε, μιλάω για το, για το 1982 που ε, μία εβδομάδα πριν παιχτεί η ταινία βλέπαμε και ένα κλιπ και βλέπαμε τον Άνω ω ως Κόναν Βάρβαρο με τα γερμανικά να, να αναφέρει καθισμένο λοιπόν στο θρονό του ότι θα κάψουμε τα ε, χωριά τους και θα βιάσουμε τις γυναίκες τους. Και γιατί αναφέρομαι στον κόσμο, γιατί ε, η σύραξη στη Συρία είναι η πέμπτη σύραξη την οποία βιώνω, αλλά είναι η μοναδική στην οποία δεν βρίσκομαι στην ίδια τη χώρα. Και όταν ακούω κάθε φορά ότι υπάρχει ε, συστηματικά λοιπόν, σεξουαλική βία η ασκείται, πάντοτε θυμάμαι αυτήν την ρίση του Άννα Φασενέγκερ, ω Κόναν ο Βάρβαρο. Και αυτό γιατί, γιατί πρόκειται για μια ιστορία που πω συμβαίνει παλιά ε, στο παρελθόν, αλλά τελικά θα μπορούσε να συμβαίνει και σήμερα, γιατί δεν έχουν αλλάξει οι τακτικέ του πολέμου. Επίση, αυτή η ρίση μα δείχνει ακριβώ ε, ε, το σε τι αναφέρεται αυτή η σεξουαλική βία, δηλαδή στο να διαλύσει τη μικρότερη μονάδα μια κοινωνία που είναι η οικογένεια. Και επίση δείχνει ότι γίνονται αλληλεπιληπτές οι γυναίκες ως ε, άτομα τα οποία δεν έχουν έναν ενεργό ρόλο, δεν λαμβάνουν αποφάσεις, δηλαδή αποτελούν απλά ένα μέλος μιας οικογένειας. Είναι η μητέρα κάποιου, είναι σύζυγο, σύζυγος ε, κάποιου, είναι κόρη ε, κάποιου. Και παρότι λοιπόν γίνονται περισσότερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας, θα πρέπει αυτές να συνδεθούν με το να δοθεί ακριβώς περισσότερη έμφαση ε, στην ενεργό συμμετοχή της, ε, των γυναικών. Και οι τελευταίες προσπάθειες ε, πραγματικά τις παρουσιάζουν μόνο ως παθητικά θύματα της επιθετικότητας των ανδρών και αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο στο πώς γίνονται αντιληπτές και σε ό,τι αφορά τον ρόλο που μπορούν να παίξουν την επίλυση των σύγκρουσεων. Και ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο τομέας της κοινωνικής βοήθειας που προσφέρει το ε, ε, ΟΗΕ. Και παρότι δηλαδή εκεί στα κλάστερς και την οργάνωση βλέπουμε ε, ότι πράγματι δίνεται περισσότερη έμφαση στο gender mainstreaming, έχουμε δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο empowerment, δηλαδή στο να λάβουν περισσότερο ακριβώς ενεργό ρόλο οι γυναίκες. Και στο ίδιο πλαίσιο ε, ε, ε, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα σεξουαλικής βίας, αλλά ε, θα πρέπει να γίνονται λεπτά και από την πλευρά των θυμάτων, από την πλευρά των γυναικών. Το 2014 τώρα η Διεθνής ε, Συνομοσπονδία για την η ε, ειρήνη και την ελευθερία προέβησε μια ε, εξέταση των σχετικών εκθέσεων και των ψηφισμάτων ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των, της βίας κατά των γυναικών στη Συρία και πραγματικά είδαμε εκεί ότι γίνονται αντιληπτές ακριβώς μόνο θύματα σεξουαλικής βίας, πράγμα το οποίο βέβαια τους αποκλεί τη δυνατότητα να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία. Η Βίνα με την υποστήριξη της, ε, του Ιδρύματος Φρίντριχ ε, Έμπερτ έχει ακριβώς ε, υποστηρίξει την, μια αντίστοιχη οργάνωση σε ό,τι αφορά την, τις διαδικασίες ειρηνευτικές, δηλαδή οικοδόμησης ειρήνης στη Συρία και με βάση τις πληροφορίες που συλλέξαμε από διάφορες οργανώσεις για την προστασία των γυναικών αλλά και από ηγέτες προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το πώς ακριβώς εργάζονται ακριβώς τις προσπάθειες, ε, τις ειρηνευτικές διαδικασίες οι γυναίκες στη Συρία, ποια είναι τα προβλήματα σε αυτή τη συμμετοχή τους και πώς η ίδια η, η διεθνής κοινότητα μπορεί να προωθεί στον εργόλο των γυναικών σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Εκεί λοιπόν η έκθεση δίνει ε, ε, έμφαση στο τι θα πρέπει να λάβει η χώρα προκειμένου να σταματήσει αυτή η σύρρηξη και το πώς μπορούν βέβαια να παίξουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο και εξωτερικοί παράγοντε. Ειδικότερα εστιάζει σε ζητήματα ε, ανάληψης περισσότερου ενεργού σημαντικού ρόλου στο οικονομικό επίπεδο, τη ε, τροποποίηση των νόμων που προβαίνουν σε δυσμενεί διακρίσει, την ε, ε, ενίσχυση τη κοινωνία των πολιτών και βέβαια την συμπερίληψη των γυναικών μέσα σε αυτή την εθνική διαδικασία. Δηλαδή περισσότερη έμφαση στην, στην ενίσχυση τη κοινωνία των πολιτών. Αλλά α δούμε λίγο περισσότερο αυτά τα ζητήματα ένα προ ένα σε ό,τι αφορά την ανάλυση περισσότερο ενεργού ρόλου στην οικονομία. Ε, Πάντοτε εστιάζουμε στη σύραξη στη Συρία, αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχει από, ταυτόχρονα μια ζωή στο επίπεδο δηλαδή, των αμάχων των, των ε, πολιτών και βέβαια οι γυναίκες ε, έχει χρειαστεί να αναλάβουν περισσότερο οικονομικό ρόλο ε, ακριβώς επειδή οι άντρες συμμετέχουν στη σύραξη πράγμα το οποίο μπορούμε να δούμε με θετικό μάτι αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια μπορεί να αποτελέσει ε, ιδιαίτερη επιβάρυνση για τις γυναίκες ειδικότερα όταν ακριβώς έχουν αναλάβει και άλλους ρόλους μέσα στην οικογένεια. Τώρα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το, το σεξ για την επιβίωση ή την, την, το ότι θα πρέπει να παντρεύουν τις ανήλικες ε, θυγατέρες τους ε, γυναίκες και άλλες τέτοιες ε, περιπτώσεις αυξάνουν την επιβάνηση για τις γυναίκες. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ευάλωτες οικογένειες μπορούν να αποτελέσουν θύματα των εκτεμιστικών οργανώσεων και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουν δηλαδή να κάνουμε τέτοιες οργανώσεις ότι δεν, έχουν, δεν εστιάζουν τόσο στις αρχές τους. Περισσότερο δηλαδή εδώ παίζουν παίζουν ρόλο ζητήματα ε, της οικονομικής κατάστασης. Βέβαια αυτό το οικονομικό empowerment ε, συνδέεται ακριβώς και με την εικόνα που έχουμε, δηλαδή ε, ε, αντίθεση μεταξύ του ρόλου των γυναικών, των ανδρών δηλαδή οι οποίοι μάχονται και των γυναικών οι οποίε είναι παθητικά θύματα. Θα πρέπει ακριβώς λοιπόν το empowerment να λάβει να, να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτό και εδώ έχουμε το παράδειγμα να αναφέρουμε τη σχετική Αφρικανική Δημοκρατία όπου είχαμε τι ε, ε γυναίκε οι οποίε συνεργάζονταν μεταξύ του στον οικονομικό φορέα ακόμα και αντίπαλων ομάδων σε μία από τι πιο αιματηρέ σειράξει που έχουμε δει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των ε, νόμων οι οποίοι προβαίνουν σε δυσμενεί διακρίσει ει βάρο των γυναικών. Σε πολλέ χώρε λοιπόν, μεταξύ αυτών και τη Συρία, ακριβώ δίνεται έμφαση στι γυναίκε ω μέλη οικογενειών και ό, όχι ω αυτόνομοι φορεί αποφάσεων. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα δίνει ε, έμφαση στην αυτονομία τους, να έχουν, ε, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν για παράδειγμα νόμοι που προβλέπουν ε, ε άνεση μισθοδοσία ή ε, οικογενειακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του να ξαναπατριστούν και όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και όπως μου είπε και μία ακτιβίστρια γίνονται λένε και πιο υπεύθυνε οι ίδιε γυναίκε για τις οικογένειέ τους, χωρίς όμως να αυξάνεται ταυτόχρονα και σε νομικό επίπεδο αυτή η ευθύνη. Επίση, ό,τι αφορά την ενίσχυση τη κοινωνία των πολιτών, έχουμε μια μεγάλη εισρωή ε, κονδυλίων και βέβαια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και εδώ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Παρ' όλα αυτά, όσοι αφορεί ε, τη κοινωνία των πολιτών και οι διεθνεί ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει που προσπαθούν να βοηθήσουν έχουν πολύ μεγάλα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, ο χώρο, τα περιθώρια λιγμών που έχουν είναι πολύ περιορισμένο. Δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικού λογαριασμού, δεν μπορούν να διαρχονται τα σύνορα εύκολα και ούτω καθεξή. Όλα αυτά θα πρέπει να να ληφθούν πολύ σοβαρά από την ε, διεθνή κοινότητα. Γιατί ουσιαστικά ε, ε, δεν επιτρέπουμε στο, στην μοναδικό δημοκρατικό θεσμό που υπάρχει ακόμα στη Συρία να λειτουργήσει σωστά. Και έλαβα ένα μήνυμα στι αρχέ του Σεπτεμβρίου από μία οργάνωση γυναικών από τη Συρία και θα ήθελα να σα διαβάσω εδώ για να αντιληφθείτε και τι συμβαίνει εκεί. Μου γράφει λοιπόν ότι αγαπητή Σάρα η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Ο Αύγουστο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Είχαμε περίπου 20 βομβαρδισμού καθημερινά. Όλα σχεδόν τα κτίρια έχουν καταστραφεί. Όλες οι ε, δραστηριότητε μα έχουν μεταφερθεί σε άλλε εγκαταστάσεις, αλλά ε, τι τελευταίε δύο εβδομάδε του Αυγούστου είχαμε ακόμα περισσότερα προβλήματα ακριβώ λόγω των βομβαρδισμών. Ε, όλοι μα είμαστε καλά, αλλά χρειάστηκε να σταματήσουμε τι δραστηριότητε μα και στις αρχές του χρόνου ο πληθυσμό εδώ ήταν 11.500 άτομα, τώρα έχουμε μείνει μόνο 500 και μόλι θα έχουμε περισσότερε πληροφορίε στη διάθεσή μα θα σε ενημερώσουμε. Ε, πολλούς χαιρετισμούς οι ε, γυναίκε τη Συρία, όπως αναφέρεται και στην έκθεση δεν επιθυμούν να χάμε τα ως ε, πιόνια. Δηλαδή, ε, συχνά δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο εκπροσωπούνται, πώς μπορούν να ποιο είναι ο αντίκτυπο ε, που έχουν στη Συρία και ουσιαστικά ε, δεν έχουν κανένα ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική διαδικασία. Όταν είχα βρεθεί στη Σομαλία το 2007, ε, ε, πρόκειτο να συναντήσω τι επιτροπέ ανδρών και γυναικών μια ενός καταπλησμού εκδιωγμένων ε, στο Βελκάγιο και ε, όταν είχαν λοιπόν συγκεντρωθεί γύρω στα 100 άτομα γύρω μου ε, και είχαν πάρει τις θέσεις του ρώτησα πού είναι η Επιτροπή των Γυναικών. Ο διερμηνέας μου προέβη στη μετάφραση και ένας άνδρας φώναξε θέλει να δει γυναίκες, φωνάξτε μια-δυο γυναίκες να έρθουν εδώ. Και βέβαια η, ο τρόπος που αντιμετωπίζει η διεθνή κοινότητα τη της, της, Συρία είναι ε, αντίστοιχη με αυτή. Δηλαδή είχα λάβει πρόσφατα ένα τηλεφώνημα από ένα ειδικό γραφείο, από μια ε, οργάνωση και κάποιο μου είπε ότι ε, θα, διαθέσουν κάποια κονδύλια για μια-δυο γυναίκε, έτσι όπω το είπαν, για να μεταβούν στη Γενέβη. κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει εδώ να ενωθούμε οι γυναίκε για να δείξουμε περισσότερο τον ρόλο που μπορούμε να παίξουμε. Μια Συριακή οργάνωση είχε κάνει και ένα σχετικό μικρό φίλμο που έδειχνε ακριβώ το πώ μπορεί η γυναίκα να βρει την γυναίκα τη, τη, τη φωνή της, να λάβει δηλαδή ένα ρόλο. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ως πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το να μην αναλαμβάνουν δράση οι γυναίκες. Όσο, όπως οι περισσότερες εκθέσεις αναφέρουν, το 75% ε, ε, αποτελούν θύματα των σύνταξεων. Οπότε αν δηλαδή προσθέσουμε ε, τον αριθμό των γυναικών με ε, τον αριθμό των ατόμων ηλικία κάτω των 18 ετών θα δούμε ότι αποτελούν την, ε, την πλειοψηφία των πληθυσμών σε οποιαδήποτε επίπεδο, είτε μιλάμε για ένοπλη σύνταξη, είτε μιλάμε για περίοδο ειρήνης. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ζητάμε το υπόλοιπο 25% του πληθυσμού να βρει μια λύση, να προβεί στην ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά η εμπειρία μα έχει δείξει ότι όταν βασιζόμαστε σε μια μειοψηφία μια κοινωνία για να προβεί στην ειρήνη, αυτή η ειρήνη θα είναι εύθραυστη, δεν θα θα λειτουργήσει καθόλου. Ε, έχουμε μάθει κάποια μαθήματα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την εθνότητα ή την θρησκεία, αλλά δεν έχουμε μάθει αυτά τα μαθήματα σε ό,τι αφορά ε, το φύλλο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε μαζί μας την αδελφή Αντζελίκ Ναμάικα, συντονίστρια τη μη κυβερνητική ε, οργάνωση ΚΡΑΤ της Λαϊκή Δημοκρατία του Κονκό, εμπειρογνώμονα προσκεκλημένη από την ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε διπλή χαρά που σας έχουμε εδώ μαζί μας, γιατί συνειδητοποιούμε τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε προκειμένου να έρθετε εδώ να μοιραστείτε μαζί μας ε, σήμερα το απόγευμα αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση. Και γι' αυτό ακριβώ ε, επιμένω ότι σας ευχαριστούμε διπλά. Ήταν τεράστια προσπάθεια που κάνατε για να μπορέσετε να είστε παρούσα εδώ σήμερα. Η Αδελφίνα Μάικα ε, βραβεύτηκε από τον ύπατο αρμοστή για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών το 2013 με το βραβείο ε, τη πρόσφυγα Νάνσεν για τα όσα έκανε στην ε, βόρεια ε, πλευρά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κανκό με εκτοπισμένες γυναίκες και γυναίκες θύματα κακοποίησης. Επιμένω ότι περιμένουμε με αναπομονησία να μας πείτε ε, όσα έχετε να μας πείτε, την εμπειρία σας και να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ μαζί μας και θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Σας ε, ε, χαιρετώ όλους και σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας ακούσετε σήμερα. Μου ζήτησαν να σας παρουσιάσω την κατάσταση και την πρόοδο των γυναικών που είναι θύματα ένοπλων σειράξεων. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι σήμερα ακόμα γίνεται λόγος για τη συμμετοχή των γυναικών ε, στην ειρηνευτική διαδικασία, στην ασφάλεια, ε, και ταυτόχρονα οι γυναίκες αυτές από τη στιγμή που γεννούν παιδιά ε, είναι αυτές οι οποίες μαθαίνουν στα παιδιά τι θα πει η ειρήνη και ε, αυτό κάνουν μέχρι να ενηλικιωθούν. Ε, καταρχάς οι γυναίκες που είναι θύματα ένοπλη σύραξη ζουν μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια. Έχουν χάσει όλα τους τα αγαθά, τον άντρα τους, τα παιδιά τους, έχουν χάσει τις σπουδέ τους, την παιδεία τους και όπως ξέρετε ε, ορισμένες φορές ε, ακόμα και έχουν καταλήξει στην πείνα γιατί όπως ξέρετε οι ένοπλες σειράξεις οδηγούν και στην πείνα. Οι γυναίκες αυτές οι οποίες ε, υποφέρουν από τραυματισμούς αναγκάζονται να ζουν και να αναζητούν τη χαρά και την ειρήνη. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες προκειμένου να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία και να αρχίσουν να μιλούν για την ειρήνη σε άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες τι οποίες έχουμε ξεκινήσει. Καταρχάς ε, ε, αλφαβητισμό για να του μάθουμε γράμματα ώστε να έχουν οι γυναίκες εφόδια να ξεπεράσουν το φόβο του. να ε, ξεπεράσουν τα, οπισθοδ... τις οπισθοδρομικές συνήθειες που λένε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να παίρνουν το λόγο. Ε, προσπαθούμε να μάθουμε σε αυτές τις γυναίκες να διαβάζουν, να γράφουν και να κάνουν αριθμητικές πράξεις. Και πρέπει να μπορούν αυτές οι γυναίκες να μιλούν και ανάμεσα στις άλλες γυναίκες, πολλό δε μάλλον ανάμεσα και σε άλλους άνδρες, ώστε να μιλήσουν για την ειρήνη. Έχουμε επίσης ε, και κάποια μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και μαθήματα ε, κοπτοραπτικής και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την τοπική κοινότητα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες γίνονται προκειμένου να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα τραύματά τους, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους και να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, να τα μορφώνουν για το τι είναι ειρήνη, ασφάλεια από τη στιγμή που γεννιούνται. Πώς μπορούν λοιπόν ε, αυτές οι γυναίκες στη συνέχεια να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ειρήνη. Οι γυναίκες αυτές αφού μάθουν γράμματα αρχίζουν να μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιες συναντήσεις. Καταρχάς στην τοπική τους κοινότητα επιτόπου και φτάνουν ορισμένες φορές να συμμετέχουν και σε πολύ μεγάλες συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκεί μιλούν ανοιχτά μιλούν στις κυβερνήσεις για την κατάσταση για την ειρήνη και χαίρομαι για το θάρρος αυτών των γυναικών που υποφέρουν, που μπορούν να μιλήσουν για αυτά τα οποία ε, τους έχουν ε, αγγίξει και τους έχουν χτυπήσει. Και μετά τι αλλάζει σε αυτές τις γυναίκες, ποια είναι η πρόοδος. Μετά από αυτή την εκπαίδευση και αυτές τις δραστηριότητες προς τις γυναίκες αρχίζουν να μπορούν να αναλαμβάνουν ε, τα ενία τη ζωή τους μόνες τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε, να φροντίζουν την υγεία των παιδιών τους, ε, την εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά και να μπορούν να τα θρέψουν. Και ε, ε, ξέρετε ότι αυτά δεν αρκούν βέβαια για αυτές τις γυναίκες, γι' αυτό και ζητήσαμε από τα δημοτικά σχολεία να δέχονται τα παιδιά τους. Έχουμε καταφέρει να χτίσουμε σχολεία, να ανοίξουμε παιδιατρικές κλινικές και καθώς επίσης θα θέλαμε να υπάρχει και με ευθύριο ώστε να μπορούν τουλάχιστον οι γυναίκες αυτές να έχουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη να δίνουν μάχη για την ειρήνη. Αν είναι πάρα πολύ στερημένες αυτές οι γυναίκες, είναι ακόμα μια ευκαιρία να βρουν ένα τρόπο ε, να μην ε, τραυματιστούν περισσότερο και να μην γίνουν πιο δυστυχισμένες. Θα σταματήσω λέγοντας ότι το θάρρος αυτών των γυναικών είναι αυτές που μου έδωσαν ε, το, την ιδέα να έχουμε αρτοπία σε βιομηχανική κλίμακα και να έχουμε και μικρές περιοχές τις οποίες μπορούν να καλλιεργούν. Ε, οι γυναίκε αυτέ είναι αυτέ οι οποίε μα πρότειναν όλε αυτέ τι λύσει. και πλέον έχουμε καταφέρει να έχουμε μια καινοτομία που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν κάποια πράγματα είναι γυναίκες οι οποίες υπήρξαν θύματα, θύματα πολέμων και που άρχισαν σιγά σιγά και άρχισαν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους και από το θάρρος που επιδεικνύουν καθημερινά. Ολοκληρώνοντας, για το μέλλον σκεπτόμαστε να έχουμε ένα σχολείο το οποίο θα είναι επιμόρφωση για όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες έχασαν τόσα χρόνια ε, και έχασαν και τα χρόνια σπουδών του ώστε να μπορέσουν ε, να έχουν τα πνευματικά εφόδια ώστε να μπορούν να αποφασίσουν μαζί με τους υπόλοιπους για την ειρήνη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες να μάθουν γραφή και ανάγνωση και να συνεχίσουν να μπορούν να ζουν ε, ε, και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ολοκληρώνοντας, να σας ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ όλους τους δωρητές από πλευράς Ευρώπης ε, που βοηθούν αυτές τις γυναίκες της χώρες μας που ε, υποφέρουν από την βία του πολέμου αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ό,τι καλύτερο για όλους. Η para και για να ολοκληρώσουμε με τις παρεμβάσεις αυτές ε, στο πρώτο πάνελ, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τζάνετ Μπένσχοφ, πρόεδρο του Global Justice Center των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπειρογνώμονα προσκεκλημένη από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Μπένσχοφ θα μας μιλήσει για την πρόεδρο και τις προκλήσεις από την έγκριση του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς ε, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συμπληρώσουμε ε, μία εικόνα ε, του τι ακριβώς κάνουν αυτές οι οργανώσεις, να ακούσουμε και τι κάνει η δική σας. Έχετε το λόγο. Thank you very... Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι, είναι για μένα μεγάλη τιμή να έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στο σώμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο, στην πρώτη γραμμή της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο φύλων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ ενώ χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες χριστιανές έχουν, συνεχίζουν να βρίσκονται εχμάλωτες και να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπόκο Χαράμ στη Συρία. Οι χριστιανές, όπως επίσης στο Ιράν και στο Ιράκ, έχουν να αντιμετωπίσουν τους εξαναγκαστικούς γάμους, βιασμούς, εξαναγκαστικές εγκυμοσύνες. Και αναρωτιέται κανείς, τι σημαίνει το ψήφισμα 1325, γιατί δεν ακολουθείται η αρχή της υποχρέωσης προστασίας. Τι νόημα είχε η δήλωση ποτέ ξανά. Όταν το Συμβούλιο ασφαλεία του ΟΗΕ ψήφισε το 1325, ακολούθησαν 7 ακόμα ψηφίσματα για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών, στα οποία αναφερόταν στην καταπολέμηση της ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στι ερευνητικέ αποστολέ. Έχει σημειωθεί πρόοδο. Αλλά όχι όσον αφορά αυτό τον σημαντικότατο στόχο συνεχίζονται οι μαζικοί βιασμοί γυναικών και κοριτσιών και να χρησιμοποιεί το βιασμό ως όπλο πολέμου στο 1 τρίτο των πολεμικών συγκρούσεων στον κόσμο σήμερα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εδώ και 15 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη και πολλά κράτη συνεργάζονται για να σταματήσει ο βιασμός ως όπλο πολέμου. Αλλά πού οφείλεται αυτή η αποτυχία μετά από 15 χρόνια δεν είναι εξαιτία της αδράνειας, είναι εξαιτία άλλων λόγων στους οποίους θέλω να αναφερθώ. Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να ψηφίσει το 1325 βασιζόταν στο κεφάλαιο του καταστατικού των Ηνωμένων ε, Εθνών που αναφέρεται στην προάσπιση της ασφάλειας και ειρήνης και ως εκ τούτου στην καταπολέμηση των σοβαρών παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου η πρώτη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβουλίο Ασφαλείας το 2002 ήταν ξεκάθαρη. Το ψήφισμα 1325 σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει ο βιασμός στις, στο πόλεμο και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εφαρμόζονται οι συνθήκες της Γενέβης και τα προαιρετικά πρωτόκολλα σε αυτές από όλα τα κράτη χωρίς διακρίσεις κατά των γυναικών. Αλλά οι ελλείψεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι απολύτως ξεκάθαρες και ορατές όταν κοιτάμε την αποτυχία του 1325. Δεν λειτουργεί. Γιατί βασίζεται, βασίζονται οι συνθήκες της Γενέβης σε ένα ιστορικό ε, παράδειγμα όπου φανταζόμαστε ε, πόλεμο μεταξύ στρατών που αποτελούνται από άντρες που χρησιμοποιούν πυρομαχικά ε, και ε, ένα μοντέλο πολέμου στο οποίο το μεγαλύτερο μέλος των θυμάτων είναι οι στρατιώτες που θα περιθαλπούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Δεν είναι έτσι οι εμπόλεμες συγκρούσεις σήμερα. Πρόκειται περισσότερο για, εσωτερικούς, για εμφύλιους πολέμους είτε για συγκρούσεις όπως εκείνες τις οποίες συμμετέχει το ISIS. Συγκρούσει στις οποίε ο άμαχο πληθυσμό και ιδιαίτερα οι γυναίκες υφίστανται εξίσου τις συνέπειες. Το 90% των απολειών στον πόλεμο σήμερα είναι άμαχοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Και η ιατρική τους περίθαλψη δίνεται σε ε, πολιτικά νοσοκομεία, όχι σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Ακόμα και το είδο των τραυματισμών είναι διαφορετική. Πρόκειται για το μόλις από τον ιό του AIDS, μετά από βιασμό, εγκυμοσύνες μετά από οι οποίες μάλιστα κυρίως αφορούν γυναίκες κάτω το 18, καταστροφή του αναπαραγωγικού συστήματος και των γενετικών οργάνων των γυναικών, το οποίο σημαίνει ότι καταστρέφεται πλήρως η υγεία, η σεξουαλική και η αναπαραγωγική της γυναίκας για το υπόλοιπο της ζωής της. Επομένως, το κάλεσμα του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου του ΕΕ αναφέρεται στις συνθήκες της Γενέβης που δεν είναι όμως κατάλληλες για την αντιμετώπιση των συμμετρικών προβλημάτων γιατί βασίζονται σε μια πατριαρχική κοινωνία και σε ένα άλλο μοντέλο πολέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτούν οι γυναίκες είναι να προστατευτούν τα δικαιώματά τους η καταπολέμηση του βιασμού ως όπλου πολέμου δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα υπόλοιπα εγκλήματα πολέμου ή η χρήση ε, όπλων μαζικής καταστροφής. Οι θάνατοι των γυναικών δεν καταμετρούνται ως απώλειες ε, πολεμικές. Οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα. Το 1325 ζητά να τερματιστεί η ατιμορρησία, αλλά για ποια εγκλήματα. Πώς ορίζονται αυτά τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά των γυναικών και των κοριτσιών, επειδή το δίκαιο έχει διαμορφωθεί μέσα από ένα ανδρικό πρίσμα, δεν αναγνωρίζονται καν ως εγκλήματα πολέμου. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι πώς θα εφαρμόσουμε το 1325, αλλά πώς θα διορθώσουμε τις ε, συνθήκες της Γενέβης, έτσι ώστε να καλύψουν και τις γυναίκες. Κανένα ψήφισμα του ΟΗΕ δεν μπορεί να σταματήσει το βιασμό ως όπλο πολέμου. Αλλά οι συνθήκες των, της Γενέβης μπορούν να διορθωθούν, έχουν τις σχετικές ε, δικλίδες τροποποίησης. Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη κάνουν ό,τι χρειάζεται, χρειαστεί, έτσι ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σέβονται κάθε πρόβλεψη των συνθηκών της Γενέβης χωρίς, διακρί, χωρίς διακρίσεις. Χωρίς διακρίσεις εξαιτίας του φύλου επίσης. Το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του τη διάσταση του φύλου και αυτό είναι μια ευθύνη της διεθνούς κοινότητας. Θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα συστηματικών διακρίσεων κατά τον γυναικών θυμάτων βιασμού ε, που, που παρά τις συνδίκες του, της Γενέβης ε, υπάρχουν, υφίστανται σήμερα. Οι συνθήκε τη Γενέβη έχουν την εξή φιλοσοφία ότι θα πρέπει να μειωθεί το αντίκτυπο του πολέμου προ, στατεύοντας τον άμαχο πληθυσμό αλλά και τους στρατιώτες και επίση απαγορεύοντα μια σειρά πολεμικών πρακτικών η θεμελιώδης αρχή από το 1864 είναι ότι όλα τα θύματα μιας εμπόλεμης σύγκρουσης και οι στρατιώτες και οι άμαχοι ότι τα θύματα αυτά όταν έχουν τραυματιστεί σε πολεμική επιχείρηση δικαιούνται ιατρική περίθαλψη και τα κράτη πρέπει να, την, να φροντίζουν να έχουν πρόσβαση τα θύματα σε αυτή την ιατρική περίθαλψη χωρίς διακρίσεις, χωρίς κανενός είδους διάκριση, είτε πρόκειται για εθνική, φιλετική ή ε, διάκριση εξαιτία του φύλου βεβαίως. Στι συνθήκε τη Γενέβη δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα, γιατί ο τρόπο αντιμετώπιση ιατρικά αυτών των περιστατικών αλλάζει καθημερινά. Ωστόσο, σε ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε εμπόλεμες περιοχές, τα θύματα των βιασμών δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έκτρωση. Οι εκτρώσεις αυτές δεν, έχει σχέση, δεν έχουν σχέση με το δικαίωμα στην έκτρωση ή με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Έχει, έχουν σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε ένα θύμα βασανιστήριων το πώ θα βοηθήσουμε μια γυναίκα που έπεσε θύμα βασανιστήριων να συνεχίσει τη ζωή της μετά. Δύο χρόνια μετά. Η έκθεση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι άρνηση παροχής πρόσβασης ε, στις εκτρώσεις για θύματα βιασμού παραβιάζει το άρθρο 13 του πρόσθετη της Γενέβης, το κοινό άρθρο 3. Είναι δύσκολο στην ανδροκρατούμενη μας κοινωνία να σκεφτεί κανείς γιατί η έκτρωση είναι ένα δικαίωμα ή κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να παρέχεται σε γυναίκες σε εμπόλεμες συγκρούσεις. και μέχρι πρόσφατα σε καμία από τις προσπάθειες εφαρμογής του 1325 δεν είχε αναφερθεί ότι ίσως τα μέτρα που χρειάζονται ε, οι γυναίκες, τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να προστατεύονται για τις γυναίκες κατά τη διόρκεια των πολεμικών συγκρούσεων διαφέρουν από εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γίνονται σεβαστά τα οποία γίνονται σεβαστά σε περίοδους ειρήνης. το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 21-22 και πρόσφατα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα στην έκτρωση για τα θέματα βιασμού. Το Ενωμένο Βασίλειο έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή αυτή τη πολιτική με την α, DFED e να δίνει τον, τη δυνατότητα στις οργανώσεις τις οποίες χρηματοδοτεί άλλο να ενημερώνει τις οργανώσεις τις οποίες χρηματοδοτεί ότι ανεξαρτήτως του εθνικού δικαίου έχουν την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση στην έκτρωση για θύματα βιασμού ε, σε, για τα θύματα πολέμου και ότι σε περίπτωση που το αρνηθούν μάλιστα αυτό μπορεί να συνιστά ε, μια ε, παραβίαση του άρθρου της Εθήκης της Γενέβης και συγκεκριμένα ε, σκληρή απάνθρωπη και μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, που είναι ο δεύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο και ορισμένα κράτη-μέλη της ακόμα περισσότερο σημαντικά, θα έπρεπε να ακολουθήσει την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν αυτό αρχίζει να εφαρμόζεται στην πράξη, θα αλλάξουν δραματικά οι συνθήκες για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο, στις εμπόλεμες περιοχές. Καμία χώρα που μόνη της ίσως να μην μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και γιατί. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιβάλει μορατόριουμ στην κατά τη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών οργανώσεων που σημαίνει ότι όταν χρηματοδοτούν τον Ερυθρό Σταυρό ή την Ερυθρά Εμισέλινο ή άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις οι Ηνωμένε Πολιτείε απαγορεύουν την παροχή πρόσβαση ε, στις εκτρώσεις. Το οποίο στην πράξη θα σήμαινε ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σπάσει αυτό το αδιέξοδο να ζητήσει τα χρήματα που παρέχει εκείνη να υπολογίζονται διαφορετικά από τα χρήματα τα οποία προέρχονται από τι ΗΠΑ και να έχουν τη δυνατότητα οι ε, οργανώσεις οργανώσει που προσφελούνται από αυτή τη βοήθεια να τα χρησιμοποιήσουν και για την παροχή εκτρώσεων για την παροχή ε, ιατρικής περίθαλψης ε, σε χώρες όπως η Νιγηρία ή η Συρία για την περιοχή ε, περίθαλψης λοιπόν στις γυναίκες και τα κορίτσια. Το 2014 το 4,77% του UNFPA προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ το 49,2% ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, η UNFPA συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή την απαγόρευση των εκτρώσεων που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το 1 τρίτο των κοριτσιών που σώθηκαν από τα χέρια του Μπόκο ήταν έγκυες. Και παρόλα αυτά, οι Ηνωμένε Πολιτείες δημοσίως δήλωσαν ότι η UNFPA δεν έχει πολιτική που να προωθεί τις εκτρώσεις ή τον οικογενειακό προγραμματισμό στην Ιγυρία. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα του βιασμού ως όπλου πολέμου. Το πιο σημαντικό πράγμα που κατάφερε η συνθήκη της Γενέβης, οι συνθήκες της Γενέβης, ήταν να σταματήσει η χρήση των παράνομων όπλων πολέμου. Γιατί τα κράτη του κόσμου φοβούνται την διεθνή κατακραυγή, όπως φάνηκε στην περίπτωση της χρήσης χημικών όπλων από τη Συρία. Το επόμενο βήμα βέβαια είναι να σκεφτούμε ότι η καταπολέμηση της τιμωρησίας ή το γεγονός ότι ε, διώχθηκαν εκείνοι που χρησιμοποίησαν παράνομα όπλα, ποτέ δεν σταμάτησε κανένα από το να χρησιμοποιήσει παράνομα όπλα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι το γεγονό ότι διώχθηκαν οι, οι, οι δράστε ε, αυτών των χημικών επιθέσεων που σταμάτησε τη χρήση των χημικών όπλων. Ήταν όταν τα κράτη συμφώνησαν μεταξύ τους ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των χημικών όπλων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει την χρήση του βιασμού όπλου πολέμου και η Διεθνής Οργάνωση Ερυθρού Σταυρού έχει εξειδικεύσει ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ο βιασμός χρησιμοποιείται ως τακτικό όπλο υπό την έννοια της συνθήκης της Γενέβης. Στη Συρία οι γυναίκες και τα κορίτσια κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τους βιασμούς από ό,τι από τα χημικά όπλα. Και η διαφορετική μεταχείριση που υφίστανται στα διάκριση. Ο βιασμός τόσο πολύ χρησιμοποιείται και έχει γίνει συνήθιση χρήση του στις εμπόλεμες περιοχές που δεν θεωρείται, που δεν φανταζόμαστε ότι, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, ως παράνομο όπλο όπως σκεφτόμαστε για παράδειγμα για τα χημικά όπλα ή για τα όπλα διασποράς στη Ρουάντα. πάνω από 250.000 γυναίκες που υπήρξαν θύματα βιασμού είτε πέθαναν είτε αργότερα εξαιτία των επιπτώσεων του βιασμού πέθαναν είτε κατά τη διάρκεια του βιασμού είτε μετά. Και αυτές οι απώλειες όμως δεν καταγράφησαν ποτέ ως απώλειες πολεμικές. Ε, κατεγράφησαν απλό και το απλώς για θάνατη ε, εξαιτία βίων περιστατικών. Δηλαδή αυ, αυτό το στοιχείο από μόνο του δείχνει την οτροπία μας. Υπάρχει, υπάρχουν κάποια στοιχεία προόδου, κάποια στοιχεία ενθαρρυντικά. Στην περσινή σύνοδο του ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας σε εμπόλεμες ε, συνθήκες, ο William Hague αναγνώρισε από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ο βιασμός είναι πάντοτε σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως όπλο, τότε είναι επιβαρυντικό στοιχείο η χρήση του. Και η πλατφόρμα του Πεκίνου ζητά ο βιασμός, η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου να προσθεθεί στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα δίωξης τέτοιων εγκλημάτων από το ποινικό δικαστηρίο. Έχουμε τώρα τις συνθήκες ε, που υπάρχουν μετά από μια πολεμική σύγκρουση. Έχουμε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της, πολιτικής, ε, της πολεμικής σύγκρουσης αλλά μετά έχουμε μια σειρά εθνικών νομικών προβλέψεων που μπορεί να υφίστανται. Το ε, δίκαιο μετά την σύγκρουση δεν αναφέρεται καν στο ανθρωπιστικό δίκαιο, δεν αναφέρεται καν στο 1325. Το ανθρωπιστικό δίκαιο έχει σχεδιαστεί με μια φιλοσοφία ανταπόκρισης, αντιμετώπισης των φρικτών εγκλημάτων που διαπράττουν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Επιτροπή ΣΥΝΤΑΟ του ΑΙΑ για τα δικαιώματα των γενικών δηλαδή έχει ε, ε, ε, δημοσιεύσει μια σειρά συμπερασμάτων που καταδεικνύουν αυτές τις διαφορετικά νομικά πλαίσια που εφαρμόζονται πριν και μετά και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να, απαντήσει, να απαιτήσει το 1325 αλλά και τις σχετικές νομικές προβλέψεις να εφαρμοστούν στην πράξη. Είναι πρωτοφανής ιστορικά η δέσμευση στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το διεθνές νομικό πλαίσιο έχει εξελιχθεί και αντεκατοπτρίζει αυτήν την πολιτική βούληση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο αναφέρεται στα εγκλήματα αυτά. Έχουν δημιουργηθεί επίσης και νέοι φορείς όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γι' αυτό ε, εγώ είμαι αισιόδοξη. Το 1325 και σχετικές νομικές προβλέψεις μπορεί να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να πάψουν να υφίστανται αυτές τις παραβιάσεις οι γυναίκες και να ε, προστατευτούν η ζωή των γυναικών και των κοριτσιών στις εμπόλεμες συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να το πράξουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας κυρία Πένσοβ. Ε, πραγματικά παρουσιάσατε μια σκληρή πραγματικότητα ε, σε πολλές πτυχές, ε, τις οποίες ε, επανειλημμένως έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα κάνετε και εσείς αλλά και οι άλλες δύο συναδελφοί σας που μίλησαν στον πρώτο γύρο ομιλητών, ε, όχι για τα όσα μας είπατε σήμερα, αλλά για τα όσα κάνετε κάθε μέρα στις ε, οργανώσεις σας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν ε, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις εργασίες μας και γι' αυτό ακριβώς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την εργασία την οποία εκπροσωπείτε εσείς σήμερα αλλά πίσω από εσά βρίσκονται Χιλιάδε άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και τώρα θα ξεκινήσει ένας ε, πρώτος γύρος συζήτηση. Ε, θα δώσουμε τον λόγο στους ευρωβουλευτές για να παρέμβουν ή για να θέσουν ερωτήσεις ή να κάνουν οποιαδήποτε παρατήρηση. Όποιος θέλει τον λόγο παρακαλώ. Η κυρία Χίμενες Πεσέρης χιμενε ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς ε, θα κάνω μια πολύ σύντομη παρέμβαση για να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας ε, τις ε, ομιλήτριες για όλες τις προσπάθειες που έκαναν για να βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας. Από αυτές τις τρεις παραμβάσεις που ακούσαμε είχαμε μια τελείως διαφορετική προοπτική από την καθεμία. Η μία αντιλαμβάνεται και βοηθά με διαφορετικό τρόπο, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Το γεγονός ότι προσπαθούμε, όπως ακούστηκε εδώ επανειλημμένως, οι γυναίκες αυτές να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να συνεχίσουν τη ζωή τους είτε ξεπερνώντας ε, ε, την ένοπλη σύραξη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι τα τραύματα όταν κάποιος είναι θύματα, διότι ε, ένα σχεδόν όλο το νομοθετικό μου έργο σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποστήριξη προς τα θύματα εγκλημάτων και κυρίως τις γυναίκες θύματα βίας λόγω και σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να σας πω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υπάρξει εκθέσεις ε, για τις γυναίκες σε και πάντα δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι πιέζουμε με τις τροπολογίες μας. Σήμερα ψηφίστηκε άλλωστε και μια έκθεση για την ε, ανάπτυξη και τις δυνατότητες ε, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που ε, βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Επίσης είχαμε και την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και εγώ ήμουνα συντάκτρια της σχετικής γνωμοδότησης και εκεί στην έκθεση αυτή γίνεται μνήα στην εξάπλωση της τρομοκρατίας και της ένοπλης ε, σύραξης στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική όπου υπήρξε ουσιαστική αύξηση της βίας και υπάρχουν βιασμοί και δουλεία γυναικών και νεαρών κοριτσιών που χρησιμοποιείται συστηματικά ως όπλο πολέμου. Επίσης υπάρχει μια παράγραφος που υπενθυμίζει τη συμμετοχή των γυναικών που είναι ζωτική σημασία σε αυτή τη διαδικασία της ε, ε ειρήνευσης και του εκδημοκρατισμού μιας χώρας. Και επίσης ε, υπενθυμίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των, γεγονό, ε, των γυναικών στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, να χρησιμοποιήσουμε τις γυναίκες εδώ με θετικό πρόσημο για την ε, ειρηνευτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες που είναι ακριβώς τα θύματα χρησιμοποιείται ο όρος ε, θύματα της τρομοκρατίας και πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν γιατί ε, ακριβώς επειδή είναι θύματα ξέρουν αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι ότι είναι κάτι παραπάνω αλλά υπάρχει κάτι επιπρόσθετο ε, και δεν είναι επειδή ακριβώς είναι θύματες αυτές θα μας πούνε τι θα κάνουμε, είναι ακριβώς το αντίθετο. Και όπως μας είπε και η αδελφή Εγγέλικα και η κυρία Μπένσκοφ, οι γυναίκες αυτές ξεπερνούν τον εαυτό τους, δεν ντρέπονται ε, για τη δυστυχία που τις βρήκε. Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες αν καταφέρουν να κάνουν κάτι για την κοινότητά τους, ε, ο κόσμος θα τη σέβεται όχι ας μια γυναίκα που βιάστηκε ή ήταν ε, σκλάβα, αλλά μια γυναίκα που κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το τραγικό συμβάν. Ε, Υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές που δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατάσταση και αυτό που έχει σημασία είναι οι εθνικές κυβερνήσεις και να πιέσουμε εμείς όχι μόνο εδώ αλλά και στις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να υπάρξει νομοθεσία και ε, τα ταξίδια των αντιπροσωπιών, εγώ το λέω συνέχεια, εδώ έχουμε και την ε, πρόεδρο της αντιπροσωπείας, ε, όταν κάνουμε λοιπόν ε, ε, αποστολές εξωτερικές, όπως κάνει και αποστολές η υπηρεσία εξωτερικές δράσεις, να φροντίζουμε να ε, τονίζονται αυτά τα ζητήματα, κυρίως σε χώρους που δεν γίνονται σεβαστές οι νομοθεσίες αυτές και δεν γίνονται σε μεστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ την κυρία Μπεστερίλη, κυρία Πιόρκ. Tack så hemskt mycket till våra inbjudna gäster. Eh, tack så hemskt mycket för att ni er Precis som min kollega sa så är detta någonting som vi i jämställdhetsutskottet men även då tillsammans med vårat, vårat eh, underskottet för tycker är oerhört viktigt. Och eh, jag tycker det känns... Όπως είπε και η συνάδελφος από την άλλη επιτροπή και εμείς θεωρούμε από τη δική μας επιτροπή εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό επίσης το ότι προβαίνουμε σε ένα διάλογο κοινό ε, μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ των διαφορετικών επιτροπών σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, δηλαδή την θέση των κοινικών στις ένοπλες σύραξεις. Νομίζω πως ούτως ή άλλως στην Ευρώπη έχουμε μια μακρά παράδοση μιλιταρισμού Ε, και η κυρία Μπένσχοφ μας είπε ότι θεωρεί πως μπορούμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο από την πλευρά δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί εδώ που θεωρούν ότι μπορούμε να δώσουμε μια στρατιωτικού χαρακτήρα απάντηση στα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει ένας ε, τέτοιος ε, μιλιταριστικός χαρακτήρας, μια τέτοια προσέγγιση απέναντι στα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια σειρά από χώρε οι οποίες έχουμε μεγάλη στρατιωτική βιομηχανία και εξάγουν εξοπλισμό. εξοπλισμό. Ε, και εμείς ε, από τη δική μας ε, οργάνωση, την Αλπίνα, παρακολουθούμε στενά το τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούνται αυτή την περίοδο και στρατιωτικές συμμαχίες, ε, γίνεται λόγος για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού και μάλιστα υπάρχει και μια έκκληση προς το Κοινοβούλιο προκειμένου να ψηφίσει ε, μια, ε, μια τέτοια ακριβώς αύξηση των κοντιλίων των κρατών μελών για στρατιωτικές δαπάνε. Αν λοιπόν θέλουμε εδώ ε, σε αυτό που συζητάμε να επιτύχουμε κάποια ε, πρόοδο, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη μιλιταριστική προσέγγιση που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη. Οι γυναίκε έχουν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ειρηνευτική διαδικασία μετά από ένοπλε συγκρούσει και θεωρώ πω και εμεί εδώ θα πρέπει να ε, γυρίσουμε στι θεμελιώδει αρχέ μα, δηλαδή και στα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. Κάτι τέτοιο ε, θα είναι πολύ ε, πιο επικοδομητικό από το να ασχολούμαστε μόνο με ε, στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα. Μετά αναφερθήκατε στο, ζήτημα του δικαιώματος μετά άμβλωση, δηλαδή ε, μετά από ε, διασμό. Ε, σίγουρα θα βρείτε εδώ πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν μαζί σα, γιατί οι γυναίκε οι οποίες πράγματι έχουν γίνει θύματα στο πλαίσιο τέτοιων σειράξεων και έχουν υποστεί διασμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πρόσβαση σε δυνατότητα άμβλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδότη στο πλαίσιο τη αναπτυξιακή βοήθεια, οπότε δεν θα πρέπει εδώ να ακολουθούμε τα όσα κάνουν οι Πολιτείε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να εμποδίσουμε τι γυναίκε σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτού του δικαιώματο που έχουν, δηλαδή του δικαιώματο στην άμπλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν εδώ να λάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Ίσως να φέρεται πω αποτελεί μόνο μια πτυχή, αλλά πραγματικά είναι αποφασιστική σημασία σε ό,τι αφορά την προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε ενόπλες σειράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπιόρκ. Ε, ολοκληρώνεται το πρώτο πάνελ. Ε, λοιπόν και θα ήθελα να ζητήσω από τις ομιλήτριές μας ε, να κατέβουν ε, στην αίθουσα και να καλέσουμε εδώ στην έδρα τους ομιλητές του δεύτερου γύρου συζήτησης για να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Muy bien, pues como vamos... Eh, λοιπόν, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε θα ξεκινήσουμε απευθείας ε, με την, ε, τους δεύτερο, το δεύτερο γύρο ομιλητών. Όπως κάναμε και προηγουμένως λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε ε, τους ομιλητές του δεύτερου πάνελ. Είμαι βέβαιη ότι θα είναι εξίσου ενδιαφέρον και θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των διαφόρων απόψεων από πλευράς διαφόρων ε, οργανώσεων και δράσεων για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε λοιπόν απευθείας ε, το λόγο στους ομιλητές. Ε, πρώτα θα παρέμβει ο ταγματάρχης Στέφαν Γιώζεφ Καμιλέρη. Είναι ε, ταγματάρχης του ε, στρατιωτικού επιτηλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ασχολείται με θέματα ισότητας των φύλων, συμμετείχε σε διάφορες ε, αποστολές στην Αλβανία, στο Κοσφοπέδιο, καθώς επίσης και στη Eurofor στη Λιβύη και στο UNAFOR στην αποστολή Αταλάντα. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας λοιπόν για να κάνετε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Ταχματάρχα για την παρουσίασή σας, ε, την παρουσία σας εδώ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριε, καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας ε, προκειμένου να παραστώ εδώ και να σας ε, ε, παρουσιάσω λίγο την, την πτυχή του στρατιωτικού επιτελείου και το στρατιωτικό σχεδιασμό ο οποίος, στον οποίο βασίζονται οι αποστολές στο πλαίσιο κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Ακούσαμε ήδη κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και την, το πρακτικό έργο το οποίο λαμβάνει η χώρα σε σχέση με τις οργανώσεις των γυναικών. Εγώ ωστόσο θα ήθελα τώρα να ε, εστιάσω λίγο περισσότερο στις ε, πρακτικές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εμείς σε επίπεδο στρατιωτικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά δηλαδή την ενσωμάτωση σε αυτό το σχεδιασμό του ψηφίσματος 1325 στην, στο, στις, στις σχεδιασμού πλαίσιο λοιπόν του εμείς εγώ είμαι το μόνο αρμόδιο άτομο σε ό,τι αφορά την ε, ενσωμάτωση ακριβώ των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ζητημάτων ε, του φίλου στην ε, διαδικασία σχεδιασμού. Ωστόσο, συμμετέχω και σε επιχειρησιακό επίπεδο, για παράδειγμα, όταν στο πλαίσιο μια νέα αποστολή δεν έχει ήδη οριστεί ένα αρμόδιο για ζητήματα φύλου και επίση συμμετέχω στον, στο επιχειρησιακό κομμάτι σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του επιχειρησιακού τμήματο. Ε, επίσης, όλοι οι υπόλοιποι ε, αρμόδιοι για τον ε, σχεδιασμό εστιάζουν και αυτοί από την πλευρά της παρότι εγώ είμαι ο μόνος αρμόδιος επαφή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι μας ε, στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης για το σχεδιασμό που λαμβάνουμε έχουμε ακριβώς γνωρίζουμε πώς να ενσωματώνουμε τις πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φύλου μέσα στην διαδικασία σχεδιασμού. Ωστόσο επιτρέψτε μου να σας αναφέρω λίγο τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Και εδώ βέβαια θα είναι πιο πρακτικές οι αναφορές που θα κάνω. Οι πολιτικές λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά ε, το, το φύλλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατ' εφαρμογή του ψηφίσματος 13-25 ε, έχουν αρχίσει να ε, έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο των ε, στατιστικών ε, θεσμικών οργάνων που έχουμε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα προσχέδια που έχουμε, τα γενικά προσχέδια σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά μας έγγραφα, στο πλαίσιο για παράδειγμα των διαδικασιών διαχείριση των αποστολών μα, αποστολών μας πάντα υπάρχουν κεφάλαια που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και την ε, μεταχείριση των φύλων, οπότε αυτά τα κεφάλαια δεν μπορούν να αγνοηθούν και θα πρέπει να ε, γίνουν αντίστοιχοι σχεδιασμοί στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού των αποστολών. Επίσης, κάτι ακόμα είναι ότι όλο το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε αποστολε και σε επιχειρήσει ε, λαμβάνει εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα του ε, φύλου, η οποία βέβαια είναι προσαρμοσμένη στην εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Αυτό αποτελεί προαποτούμενο για τη συμμετοχή αυτού του προσωπικού στι επιχειρήσει και επίση ε, τα στρατηγία, δίνεται εντολή στα στρατηγία να παρέχουν επανεκπαίδευση και να διαθέτουν και κώδικες διοντολογίες σε έντυπη μορφή στα μέλη. Και αυτός ο κώδικα διοντολογία, βέβαια παρότι δεν αποτελεί νομικό κείμενο ε, αποτελεί έναν, ε, μια ηθική πηξίδα αν θέλετε διοντολογία σε ό,τι αφορά όλο το προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρήσεις. Κάτι ακόμα είναι ότι όλες οι 7 δηλαδή ε, επιχειρησιακές αποστολές ε, και επιχειρήσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή έχουν έναν σύμβουλο για θέματα φύλου ή τουλάχιστον ένα σημείο επαφή για αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η θέση δεν είναι πλήρους απασχόληση, δηλαδή δεν ασχολείται μόνο με αυτό ο σύμβουλος, αντιθέτως είναι και νομικός σύμβουλος. Πράγμα βέβαια το οποίο δεν είναι μια ιδανική κατάσταση αλλά αποτελεί ένα βήμα προς τα μπροστά. Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό ε, ε, στοιχείο είναι ότι μη επιχειρησιακού χαρακτήρα αποστολέ μα, εκπαιδευτικέ δηλαδή αποστολέ, ε, προσφέρουν εκπαίδευση στους, στο προσωπικό στι εκάστοτε περιοχέ, που σημαίνει ότι προσφέρουν και αντίστοιχη εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το φύλλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια έχουν προσαρμοστεί και στου εκάστοτε εντόπιους πληθυσμού. Η ε, αξιωματούχοι σε αυτές τις χώρες λαμβάνουν ε, πιο εντατική εκπαίδευση ενώ το κανονικό προσωπικό ε, λαμβάνει την κανονική εκπαίδευση και βέβαια και αυτού του είδους η εκπαίδευση δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα μεταχείριση των φύλων αποτελεί προαπαιτούμενο σε ό,τι αφορά την παροχή ή τη λήψη περαιτέρω εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τα, τα, στρατιωτικά ζητήματα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τα όσα συμβαίνουν επιτόπου σας είπα ότι έχουμε 7 τρέχουσες αποστολές ε, και ε, επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι τρεις είναι επιχειρησιακού χαρακτήρα και οι υπόλοιπε είναι μη επιχειρησιακού, δηλαδή δημιουργία δυνατοτήτων, ε, εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Και από γεωγραφικής άποψης Όλε δηλαδή εκτός από μία, οι έξι δηλαδή, ε, βρίσκονται ε, ε, κοντά ή πάνω στην Αφρικανική Ήπειρο. Στις περισσότερες περιπτώσει, βέβαια αυτές οι επιχειρήσεις είναι πολύ περιορισμένες σε ό,τι αφορά τον αριθμό δηλαδή των ατόμων επιτόπου, σε ό,τι αφορά δηλαδή την, την αποστολή στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Έχουμε μόνο 10 άτομα επιτόπου γιατί πλησιάζει και προ το τέλο τη προ το τέλο τη σχετική εντολή για αυτή την επιχείρηση. Ενώ από την, από την άλλη πλευρά έχουμε τι ε, ναυτιλιακέ επιχειρήσει ε, στα παράλια τη Σομαλία και στα παράλια τη Λιβύη με 900 συνολικά άτομα. Ε, αυτά, σε αυτές ακριβώς περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε η σεξουαλική βία ε, και η κακοποίηση ε, υπάρχουν ε, σε διάφορα επίπεδα και μερικές φορές η κατατόπους νομοθεσία δεν προβλέπει την προστασία των γυναικών. Για παράδειγμα στη Σομαλία δεν υπάρχουν νόμοι κατά της οικιακής βίας, της βίας στις οικογένειες ενώ στο Μαλή υπάρχει ένας υπουργό για τα ζητήματα των γυναικών αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία. Στη Λιβύη από την άλλη πλευρά υπάρχει κάποια νομοθεσία αλλά υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις ε, σεξουαλικής κακοποίησης και βίας ε, δεν κοινοποιούνται στις αρχές γιατί ακριβώς υπάρχει μια κουλτούρα ατιμορρησίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εντοπίζονται οι επιχειρήσεις μας να πω ότι σε πλαίσιο όλων αυτών των αποστολών έχουμε μία εστίαση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του φύλου, χωρίς όμως αυτή η εστίαση να είναι εκτεταμένη. Η εκπαιδευτικές ε, επιχειρήσεις έχουν πολύ μακροπιότερο αντίκτυπο ε, στου ε, στους τοπικούς ε, πληθυσμούς γιατί ακριβώς παρέχουμε σχετική εκπαίδευση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αισθήματα του φίλου σε χιλιάδες προσωπικό. Και ταυτόχρονα ο αντίκτυπο τον οποίο έχουμε δεν είναι μόνο σε επίπεδο εκπαίδευση, γιατί ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των γυναικών στι εθνικέ ένοπλε δυνάμει. Για παράδειγμα, στις, στα στρατιωτικά σεμινάρια τη Σομαλία έχουμε δει έναν αυξανόμενο αριθμό συμμετοχών ω γυναίκε δηλαδή σε αυτέ τι ε, δυνάμεις ε, ε, και ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο αυτών των στρατιωτικών σεμιναρίων είναι ήδη γυναίκες. Ποιε είναι όμως οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερις βασικέ προκλήσει, βέβαια, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλε. Καταρχήν, δεν υπάρχει ισορροπία, ισόρροπη εξορρόπηση των φύλων σε ό,τι αφορά τι ίδιε τι επιχειρήσει. Δεν υπάρχουν επιχειρησιακέ κατευθυντήρε γραμμέ, δεν υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρογνωμοσύνη και επίση δεν υπάρχει η κατάλληλη συγκέντρωση γνώσεων ε, λόγω τη διάρκεια ε, των αποστολών. Σε ό,τι αφορά την ε, ισόρροπη εξορρόπηση των δύο φίλων σε όλε τι ένοπλε δυνάμει στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι δεν ε, έχουμε φτάσει εκεί που, θα, ε, εκεί που πρέπει και βέβαια καθώς κάτι τέτοιο ισχύει στις ένοπλες δυνάμεις των, ε, ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό απηχείται αντίστοιχα και στην σύνθεση ε, των αποστολών και των επιχειρήσεων. Εάν δούμε για παράδειγμα το τι συμβαίνει σε άλλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο CPCC, εκεί η εκπροσώπηση είναι 20 έως 25% ενώ σε στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεων με βάση ανεπίσημα στοιχεία ε, το αντίστοιχο ποσοστό των, τον γενικών δηλαδή βρίσκεται στο 3 με 7%. Ε, επίσης μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ε, διοικητές ε, αποστολές κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ενώ σε επίπεδο μη στρατιωτικών τέτοιων αποστολών είχαμε δύο ε, επικεφαλής αποστολών και δύο αναπληρωτές επικεφαλής. κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι σε ό,τι αφορά αυτή την ανισόρροπη εξορρόπηση ότι ακριβώς επειδή δεν βλέπουν να ότι οι, οι τοπικέ κοινότητε λαμβάνουν ένα λαθασμένο μήνυμα γιατί δεν υπάρχει επαρχής εξορρόπηση των γυναικών στι δικέ μα ενόπλε δυνάμει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι επιχειρησιακέ κατευθυντήριε γραμμέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοιε κατευθυντήριε γραμμέ ε, σε ό,τι αφορά του τους, ε, ε, συμβούλου. δεν υπάρχει κάτι δηλαδή σε επιχειρησιακό επίπεδο και βάσει μια μελέτη baseline που κάνουμε, δηλαδή μια βασική γενική μελέτη στην οποία θα αναφερθώ, θεωρούμε πως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα βασικά θεμέλια ε, για την εκπόνηση τέτοιων επιχειρησιακών κατευθυντηρίων γραμμών. Σε ό,τι αφορά τώρα την έλλειψη του ανθρωπίνου δυναμικού και της ε, εμπειρογνωμοσύνης, ε, αυτό αφορά γενικότερα βέβαια το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούμε και μέσω αυτής της μελέτης που μόλις τώρα ανέφερα να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ένα εγγενές πρόβλημα είναι η διάρκεια των ε, ε, επιχειρήσεων, δηλαδή ο ρυθμός της ε, εναλλαγής των, του προσωπικού που συμμετέχει σε αυτές, δηλαδή 4-6 μήνες που συμμετέχουν, σημαίνει ότι οι γνώσεις τις οποίες αποκτούν χάνονται και αυτό ισχύει και για τον σύμβουλο σε ό,τι αφορά τις, τα ζητήματα φύλου του στρατιωτικού επιτελείου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ αναφερόμενος στο non-paper 20 μελών σε ό,τι αφορά την, το φύλλο, την ειρήνη και την ασφάλεια στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας ε, και άμυνας. Ε, εδώ αναφέρονται μία σειρά αποζητήματα από τα 20 κράτη-μέλη τα οποία παρουσίασαν από κενού του ανλόγου έγγραφου προκειμένου να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να διατυπώσουν μια στρατηγική. Ε, εδώ αναφέρεται για παράδειγμα το ζήτημα τη καλύτερη ε, ενσωμάτωση των ε, ζητημάτων του φύλου στο στρατηγικό σχεδιασμό και επίση την ιδιαίτερη προοπτική, την αυξημένη προοπτική του φύλου στι εντολέ των επιχειρήσεων δηλαδή τη πολιτική ασφαλεία, καλύτερε συγκριτικέ αξιολογήσει και καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη για ζητήματα ε, ε, ε, φύλων. Επίσης προτείνεται ότι θα πρέπει να λάβει η χώρα μια βασική μελέτη για την αξιολόγηση της πρόοδου που έχει επιτευχθεί και γι' αυτό και το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης κρίσεων και σχεδιασμού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση μιας βασικής γενικής μελέτης προκειμένου να αξιολογηθεί ε, η σημερινή κατάσταση ό,τι αφορά την ε, ενσωμάτωση της επιτυχή ε, του φίλου στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή από το πολιτικό στρατηγικό επίπεδο έως και το επιχειρησιακό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώ λέμε ότι είναι γενική μελέτη το στρατιωτικό επιτελείο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει και στην Task Force για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ε, φύλλο ε, ε, σε συνεργασία και με την EAS ε, και με, την, ε, με το ε, Κολέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα έχουν ξεκινήσει ήδη τις εργασίες τους για την εκπόνηση αυτής της μελέτης και αναμένουμε πως τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα ως τα τέλη του 2015. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται, υποστηρίζεται από την Ακαδημία, την Σουηδική Ακαδημία Φόλου Περνατώδη, η οποία προετοιμάζει workshop, ευθετικά workshop στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σχεδιασμού της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και ε, θα ε, συμμετάσχει ε, υποστηρικτικά και στην διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών στο επιχειρησιακό επίπεδο. Με βάση λοιπόν αυτό το κοινό non-paper των κρατών μελών και καθώς έχουμε και την επέτειο, τη 15η επέτειο του ψηφίσματος 1325, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να, ε, ε, έχουμε, να επιτύχουμε άλλα σημαντικά βήματα ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, ακριβώς τον όσο προβλέπει το ψήφισμα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σκεπτικό μας, αλλά και σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε εμείς επί τόπου. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε όλοι όσοι εργαζόμαστε σε αυτό το τομέα, δηλαδή του, του φίλου και στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Χαιρόμαστε που ένα πρόσωπο όπω η κυρία Μαρινάκη έχει αναλάβει ε, τα καθήκοντα του κύριου συμβούλου ε, για αυτό το ζήτημα στην υπηρεσία εξωτερική δράση και ε, θεωρούμε πω με αυτόν τον τρόπο θα λάβει μία ακόμα όθηση η γενικότερη ατζέντα των, του συστήματο των δύο φίλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμιλέρη ουσιαστικά μας κάνετε και εισαγωγή για την επόμενη προσκεκλημένη μας ε, που θα μιλήσει εδώ στο πάνελ η πρέσβυρα κυρία Μάρα Μαρινάκη, αρμόδια σε θέματα φύλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ευχαριστούμε για τη σημερινή της παρουσία εδώ μαζί μας και της δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρίες Πρόεδροι, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα και πολύ επίκαιρη στιγμή ε, για το θέμα που συζητούμε στα πλαίσια της επαιτίου ε, του ψηφίσματος 1325 που σημειώνει ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στην ιστορία των γυναικών, στην ασφάλεια και στην ειρήνη όπως αναγνωρίζονται στη διεθνή κοινότητα στο υψηλότερο επίπεδο από το Συμβουλίο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και πράγματι το γεγονό ότι επιλέξατε τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, διότι ε, ήταν προσπάθεια να έρθω από τη Νέα Υόρκη σήμερα το πρωί, ε, από τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες δύο μέρες και ε, πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, για τον Οκτώβριο. Ο κύριος Μαριάνο Ραχόη, ε, προείδρευσε σε μια ειδική ανοιχτή συζήτηση για τη 15η επέτειο του 1325 και σημειώθηκε εκεί ένα νέο ρεκόρ 111 ομιλητές ε, εκπρόσωποι ψηλού επίπεδου έλαβαν το λόγο για να εκφράσουν τη δέσμευσή τους ε, για τις γυναίκες στην ε, ειρήνη και στην ασφάλεια και εγώ είχα την τιμή να ομιλώ εκεί εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή μου την ιδιότητα λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον αγαπητό συνάδελφο Στεφάν Καμιλέρη αλλά και όλους εσάς διότι είναι η πρώτη ευκαιρία να συστηθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το νέο μου ρόλο ως ε, ε, επικεφαλή σύμβουλο για, για θέματα φύλου ε, για το 1325. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ στενά μαζί σας ε, και με την προηγούμενη ιδιότητα ως Γενική Διευθύντρια για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φύλου και διεθνών οργανώσεων και διαπιστώνω ότι πλέον υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση στα Ηνωμένα Έθνη αλλά ε, και ιδιαίτερη ευαισθησία και ταχεία αντίδραση από πλευράς ε, υπάτης εκπροσώπου και αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Μογκερίνη με την ε, ε, δημιουργία αυτής της νέας θέσης και το διορισμό μου για να επικεντρωθούμε κυρίως σε θέματα φύλου και στο ψήφισμα 1325 με εντολή να συνεισφέρουμε ε, στο να δοθεί προτεραιότητα το θέμα των γυναικών ε, στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ειρήνης και ασφαλείας και να ενισχύσουμε και την προβολή της ουσιαστικής δραστηριότητας που έχουμε για όλα τα σχετικά θέματα ε, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέροντας και βοηθώντας την εσωτερικό συντονισμό σε θέματα φύλων και ε, ισότητας. Ε, ε, θα υπάρχει λοιπόν συνεργασία και προσβλέπω στην πολύτιμη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια συνέπεια στην πολιτική μα και στην προσέγγιση του κόσμου, ε, το μήνυμα που θέλει να αποστείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ω πρωτοπόρο σε όλε αυτέ τι πολιτικέ και για άλλη μια φορά θα πρέπει να αντανακλώνται όλα αυτά και στις ε, πολιτικές μας. Αναφέρθηκα σε όλα αυτά στην ανοιχτή συζήτηση στη Νέα Υόρκη. Αυτό το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα ε, είναι το γεγονός ότι σίγουρα ήταν το πιο περιζήτητο ε, γεγονός, η πιο περιζήτητη εκδήλωση και καταφέραμε να έχουμε ολοκλήρωση της εκδήλωσης αυτής με ένα νέο ψήφισμα ένα ψήφισμα το οποίο είναι αναβαθμισμένο, είναι μια ε, αναθεωρημένη εκδοχή του 1325 με πολλές ε, συστάσεις οι οποίες ε, έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο μέλλον και επισέρχονται σε πολύ πιο συγκεκριμένους τομείς στους οποίους αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες. Περιλαμβάνεται το θέμα της λογοδοσίας, της ευθύνης ε, για τον κατάλληλο χειρισμό σε θέματα βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς επίσης και την ε, ε, προσφυγή στη δικαιοσύνη για να καταδικαστούν τα θύματα ανεξάρτητα της καταγωγής τους και αυτό είναι ένα θαραλέο νέο βήμα που έχει αναλάβει πλέον η διεθνής κοινή γνώμη ε, καθώς επίσης υπήρχε και μία σειρά ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στον ε, ε, αρμόδιο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, για να προστατεύει ε, σε συγκεκριμένους όρους και αναμένεται να τηρήσει μια πολύ σημαντική σειρά από δεσμεύσεις τις οποίες προσωπικά δέχτηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ασπάστηκε τις ε, ε, ιδέες αυτές όταν παρουσίασε την επίσημη έναρξη της ε, παγκόσμιας μελέτης εχθές, η οποία ε, ολοκληρώθηκε από την ε, ομάδα του Ραντίκα Κομαρσβάνη και είχε έναν από τους κύριους συνομιλητές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε πολύ μεγάλη συνεισφορά από πλευρά μα ε, και τα πάντα, ό,τι προτείναμε, έγινε αποδεκτό. The new resolution, resolution 22. Το νέο ψήφισμα, το 2242, ανοίγει το δρόμο για την επόμενη 15 ετία, ώστε να ενισχύσουμε τη, τη διάσταση του φύλου στην ειρήνη και στην ασφάλεια, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη των ΗΕ Εθνών και τις διεθνείς οργανώσεις να αναπτύξουν πιο συγκεκριμένα μέσα για τις γυναίκες στην ασφάλεια και την ειρήνη και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας, της ειρήνης ε, και των γυναικών ως κάτι θετικό το οποίο μπορούν ε, να συνεισφέρουν οι γυναίκες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των εξτρεμιστικών φαινομένων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συγκεκριμένες ποιότητε είχε το ψήφισμα 1325 όταν εγκρίθηκε το 2000. Η Ναμίμπια είχε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ε, στις 21 Οκτωβρίου όταν εγκρίθηκε και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες ε, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα συγκεκριμένα. Ε, ουσιαστικές ε, προσπάθειες μέσω πολιτικών, προγράμματων δράσης, ε, κατευθυντηρίων γραμμών, συγκεκριμένης εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Έχουν γίνει αρκετά, αλλά σίγουρα δεν αρκούν. Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν πολύ εύγλωτα στην έλλειψη απόδοσης, κάτι το οποίο δεν ε, ε, επισημάθηκε αρκετά και είναι πολύ σημαντικό, ε, αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στο επίπεδο λήψης αποφάσεων και την συμμετοχή τους κατά τη διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων. Πρόκειται για τα σημεία στα οποία μέχρι τώρα έχει αποτύχει το 1325 γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ένα ισχυρό διεθνές μέσο είναι επιτυχές ε, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να το εφαρμόσουν ε, επιτυγχάνουν. Και επομένως το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το 1325, είτε οι θύνοντες που δεν κατάφεραν να κάνουν το 1325 το κατάλληλο όχημο για να συμπεριληφθούν οι γυναίκες στην ε, διαδικασία ειρήνης και ασφάλεια με σπάνιες εξαιρέσεις που έχονται να επιβεβαιώσουν τον κανόνα όπως έγινε με την Κολομβία και τις Φιλιππίνες όπου υπήρχε συμμετοχή των γυναικών. Στη Συρία υπάρχει μια καταφανής ε, περίπτωση πλήρους αποκλεισμού των γυναικών Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις ε, μαζί τους στη Νέα Υόρκη στη ε, διάρκεια της Υπουργικής Εβδομάδας το Σεπτέμβριο και ε, εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι κανείς δεν έτεινε ευήκονους στα όσα είχαν να πούν, πολλό δε μάλλον δεν τις συμπεριλάμβανε στις επίσημες διαπραγματεύσεις. Αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε και η διεθνής κοινότητα έχει και αυτή μερίδιο ευθύνη. Πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη ε, να αναλάβουν ε, ε, τις ευθύνες τους και ο Στεφάν Μιστούρα δεσμεύτηκε ότι θα βελτιώσει τα πράγματα. Τελεία και παύλα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο γιατί δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου οι γυναίκες μέχρι τούδε, επομένως πρέπει να υπάρξει κάποια αρχή. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί έχουμε ήδη δεσμευτεί πάρα πολύ. Δεν θα επισέλθουμε σε λεπτομέρειε, διότι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη σε αυτό θέλω απλώς να πω ότι στα πλαίσια της ε, συνολικής προσέγγισης που έχουμε για την εφαρμογή του ε, ψηφίσματος 1325 ε, και του 1820, ήδη το 2008 προωθήσαμε μια σειρά από δράσεις και έχουμε συμπεριλάβει, έχουμε ενισχύσει και έχουμε εμβαθύνει στις δράσεις αυτές με βάση και τα διδάγματα που αντλήσαμε από την εφαρμογή τους. Και η προσέγγιση μας σαφέστατα είναι προς την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, ε, στο πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε ώστε να μην ε, γίνουν θύματα, ε, να μπορέσουν να επιβιώσουν σε καταστάσεις ένοπλης σύραξης και πώς μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματική δράση σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και ειρηνευτικής διαδικασίας. Και σε αυτά θα επικεντρωθούμε περισσότερο τους επόμενους μήνες. Ε, προωθούμε σίγουρα την συμμετοχή των γενικών στη διαδικασία διαμεσολάβησης και στην ειρηνευτική διαδικασία και βεβαίως ε, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές βελτιώσεις. Υπάρχει περιθώριο ε, βελτιώσεων Δεσμευόμαστε επίσης και ε, για τις αποστολές ε, διαχείρισης κρίσεων και για την κατάρτιση. Ήδη έχουμε αναλάβει την κατάρτιση των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι έχει σχέση με το φύλλο και ε, τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως τους πλέον κατάλληλους ε, να αναλάβουν αυτές τις καταρτήσεις ε, και επομένως έχουμε αναλάβει την γενικότερη κατάρτιση όχι μόνο για τις ειρηνευτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τις ειρηνευτικές δυνάμεις ε, άλλων χωρών και έχουμε και συγκεκριμένα αιτήματα από χώρες για να υπάρξει αυτή η επιμόρφωση και κατάρτιση αλλά επίσης πρέπει να εφαρμόσουμε και τα εθνικά προγράμματα δράσης για τις γυναίκες, στην ειρήνη και την ασφάλεια. Από τις 193 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών, 48 μόνον έχουν εθνικά σχέδια δράσης για την ειρήνη, ε, την ασφάλεια και τις ε, ε, γυναίκες. Τα 22 βέβαια είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε μεν και αυτό, αλλά δεν αρκεί αυτός ο πενιχρός αριθμός. Πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να προσεγγίσουμε ε, ε, με εντατικό τρόπο και τους υπολείπους ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Όσον αφορά τα κενά ε, που διαπιστώθηκαν στα πλαίσια της εφαρμογής υπάρχουν τέσσερα στοιχεία του 1325, τα τέσσερα πιπ στα αγγλικά, προστασία, συμμετοχή και πρόληψη ε, και ειρήνη. Και στον τομέα της πρόληψης ε, πάσχουμε, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια πολύ σύντομη περίληψη να πω ότι έχουμε ήδη διαθέσει 100 εκατομμύρια για πλήρη οικονομική στήριξη για θέματα ισότητας των φύλων σε γυναίκες ε, και νεαρά κορίτσια και την ενίσχυσή τους και φυσικά έχουμε συμπεριλάβει και τη διάσταση του φύλου στα πλαίσια της συνεργασίας στο μέσο ε, σταθερότητας και ειρήνης και τέλος ε, βεβαίως και θα συνεχίσει η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη αλλά ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα στην προστασία των ε, γυναικών που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως σε περιοχές τις οποίες σοβούν ενόπλες σειράξεις. Ε, ολοκληρώνοντας ε, να πω ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το ρόλο της ε, ότι πρέπει δηλαδή να μιλούμε εξ ονόματος των ε, εκατομμυρίων γυναικών και κοριτσιών που δεν έχουν οι ίδιες τρόπο να μιλήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρινάκη από τις εξηγήσεις που μας δώσατε με τις οποίες συμφωνώ 100% όταν αναφερθήκατε στην παρουσία του Προέδρου της ε, Ισπανικής Κυβέρνησης, του κυρίου Ραχόη, ε, ο οποίος προείδρευε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση ε, και να πω ότι εμείς ζητούμε όχι μόνο πράξεις, χειρονομίες μάλλον, καλής θέλησης, αλλά πραγματικότητα. Και πραγματικότητα σημαίνει ασκώ την πολιτική και ε, διαθέτω κονδύλια στον προπολογισμό και μετά από πέντε χρόνια πολύ σημαντικών εργασιών ε, κινδυνεύει να εξαφανιστεί το Ινστιτούτο για τα θέματα ισότητας των φύλων όλων ε, μετά από τα ΕΣΑ έκανε λόγω έλλειψη προπολογισμού. Επομένω, πρέπει να προωθούμε θέματα Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζουμε και με πολιτικέ και με προπολογισμό, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνονται και κατάλληλε δράσει. Να ολοκληρώσουμε με την τελευταία ομιλήτρια. Εξίσου φυσικά σημαντική με τους υπολείπους, η κυρία Ντάγμαρ Σούμαχερ, Διευθύντρια του Γραφείου των Βρυξελών ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα θέματα γυναικών, με την οποία συνεργαζόμαστε στενά, ε, συνεργαζόμαστε σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και για το καθημερινό έργο του Γραφείου και για το πνεύμα συνεργασίας ε, με ε, το οποίο πνεύμα ήρθε και να συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια και εσά και τις άλλες δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πράγματι όπως και η κυρία Μαρινάκη είπε οργανώνουν σε μια πολύ κέρια στιγμή αυτή την εκδήλωση, αυτή ακρόαση. Θα και πάλι να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια κυρία Μαρινάκη από την πλευρά της UN Women. Ε, είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που θα έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε να, ε, στα νέα, και από τα νέα σας καθήκοντα να συνεργαζόμαστε μαζί. Καλή επιτυχία λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσω παραθέτοντας τα λόγια της εκτελεστικής μας διευθύντριας, αυτό που είπε αυτή την εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι συνοψίζεται όλο το ζήτημα το εργαλείο που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου, είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να πετύχουμε πραγματικά την ειρήνευση, είναι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. Νομίζω όλοι συμφωνούμε, το ζήτημα είναι πώς θα το εφαρμόσουμε στην πράξη. Θα προσπαθήσω να, να κατευθύνω τη συζήτησή μας προς το τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο, ε, σε μια πιο ε, οικουμενική προσέγγιση, έχει υιοθετηθεί πρόσφατα ε, και στο πλαίσιο της ατζέντα για τη βιώσιμη ε, ανάπτυξη ή συμμετοχή των γυναικών ε, ως στόχος για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς επίσης και η, ε, το να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση του φύλου στην αναπτυξιακή πολιτική. Είναι σημαντικό και αυτό να μην το ξεχνούμε. Κατά το, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών έχουμε οργανώσει μια εκδήλωση Global Leaders στις 27 Σεπτεμβρίου στην οποία προσκαλέθηκαν ζητήθηκε μάλλον από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ε, εκφράσουν δημοσίως τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων και η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Ε, ποτέ άλλοτε δεν είχαν παρευρεθεί και δεν είχαν εκπροσωπηθεί ε, σε τόσο μεγάλους αριθμός αρχικών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ο Επιτροπός Τίμερμανς τώρα βρέθηκε εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν φεμινιστής και αυτό δημιούργησε μια εφορία. Όλε λοιπόν αυτέ οι δημόσιε δηλώσει των κρατών αφορούσαν το ρόλο του γυναικών όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλεία επευκαιρία τη 15η επαιτίου από την, ε, το ψήφισμα 1325. Θα ήθελα να σα ζητήσω να την διαβάσετε και μπορεί επίση να συμβολευτείτε και την ε, μελέτη, την Global Study, με τίτλο προ... Ε, Παγκόσμια μελέτη για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 στην οποία αναφέρεται στις προκλήσεις και στις συγκεκριμένες συστάσεις για τις οποίες θα μιλήσω αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση ακούγοντας και την ε, ξεκάθαρη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα αυτά για την οποία θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ο ΟΗΕ έχει οργανώσει τρεις υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις αναθεώρησης και εξετάτησης της κατάστασης. Η πρώτη αφορούσε τις ειρηνευτικές διαδικασίες του ΟΗΕ και ε, το ζήτημα των ειρηνευτικών ε, επιχειρήσεων και επίσης το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην πρόγραμμα ειρήνης και ασφάλειας. Και σε όλα αυτά τονίστηκε η σημασία του ρόλου των γυναικών. Όσον αφορά τώρα παγκόσμια μελέτη για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325, είναι ένα έγγραφο που έχει συμπτύξει ε, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δείχνει με ποιον τρόπο η συμμετοχή των γυναικών μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, της ειρήνης, της ασφάλειας, μπορεί να βοηθήσει τις ειρωνιστικές ε, διαδικασίες, μπορεί να συμβάλλει στην ανθρωπιστική βοήθεια, να καταπολεμήσει τον βίο εξτρεμισμό. Είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της μελέτης αυτής το οποίο αναφέραμε. Δίνεται μεγάλη έμφαση επίσης στη σημασία που έχει να λειτουργούν οι γυναίκες και ως ηγέτες. Κάτι που βοηθάει και την ανθρωπιστική βοήθεια και τις ειρηνευτικές διαδικασίες και την σύναψη ειρηνευτικών συνεφιών, συμφωνιών και την οικονομική ανάκαμψη και ανασυγκρότηση μιας χώρας μετά από ένα πόλεμο. Αυτά δεν είναι μόνο λόγια, σχήματα ρητορικά, έχουμε και στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σημασία του συμμετοχής των γυναικών. Ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει από την μελέτη και αναφέρεται και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα με μεγάλη έλλειψη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην ειρήνη και την ασφάλεια είναι η έλλειψη χρηματοδότησης προς οργανώσεις γυναικών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οι απερώτητοι πόροι. Γι' αυτό θα ήθελα να ανακοινώσω ότι θα δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο Global Acceleration λέγεται από την πλευρά του ΟΗΕ που θα χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτούνται οι οργανώσεις εκείνες των γυναικών που ασχολούνται με την ειρήνευση και με την ανθρωπιστική βοήθεια. Κάποιες από τις συστάσεις της παγκόσμιας μελέτης Ποτέ δεν θα πρέπει να διοργανώνονται ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή γυναικών. Θα πρέπει να τους δίνονται κίνητρα και οικονομικά δυνατόν, έτσι ώστε να συμμετέχουν και οι γυναίκες ενεργά, όχι απλώς ως παρατηρητές στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το 15% των πόρων που δίνεται για μια ανασυγκρότηση μετά από πόλεμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Θυσμικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται επίσης στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι καθώς επίσης και τη δημιουργία ενός άτυπου συμβουλίου επιρρογνωμόνων για την ισότητα των δύο φύλων, έτσι ώστε ε, οι πληροφορίε και τα στοιχεία από την κοινωνία των πολιτών να φτάνουν στο Συμβούλιο Ασφαλεία πιο συχνά. Θα πρέπει επίση να, να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στι ειρηνευτικέ δυνάμει, στι δυνάμει των κυανοκράνων ή δυνατόν και με οικονομικά κίνητρα. Η το κατά πόσον έγινε σεβαστή η υποχρέωση συμμετοχή των γυναικών θα πρέπει να είναι ένα από τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη των ε, υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ΟΕΕ. Καθώς θα, θα, θα, πρέπει επίσης να ε, γίνονται έρευνες αμέσω, μόλις υπάρχουν καταγγελίες για παραβιάσει των δικαιωμάτων των γυναικών από τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Ε, βλέπω ότι δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, οπότε δεν θα μιλήσω και πολύ περισσότερο όσον αφορά την ε, έκθεση και, ε, και το ψήφισμα και τι συστάσει σχετικέ με το ψήφισμα. Θα ήθελα να σα ζητήσω να, να τι διαβάσετε στην έκθεση. Σα ευχαριστούμε. Η συμπρόεδρο έπρεπε να φύγει από την αίθουσα γιατί έπρεπε να προλάβει την πτήση τη. Γι' αυτό θα συνεχίσω εγώ να προεδρεύω τι συνάντησει μα, τι ακροάσει μα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη του Κοινοβουλίου, στους βουλευτές, αφού ευχαριστήσω τους ομιλητές μας. Και τον Ταγματάρχη Καμιλέρη και τις δύο πρέζες. Ας ε, κάνουμε μια μικρή συζήτηση. Κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, καθώς εδώ έχουμε να κάνουμε με το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών σε ένοπλες σειράξεις. Ε, πραγματικά ε, ήταν σοκαριστικά τα όσα ακούσαμε και με άγγιξαν Και βέβαια ε, με εκπλήσει το γεγονό ότι συχνά δεν μιλάμε για τι ε, γυναίκε στη Συρία οι οποίε ε, τελικά είναι αφημένε στι δικέ του δυνάμει, το να επιβιώσουν μόνε του. Δηλαδή μιλάμε για ένα σωρό διασκέψει, για συναντήσει και ούτω καθεξή, αλλά δεν μιλάμε για τι γυναίκε στη Συρία. Ακούμε για μασικού βιασμού κοριτσιών και γυναικών στη Συρία και αν όλα αυτά συμβαίνουν τότε θα πρέπει να αναλάβουμε εκτάκτω δράση. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πιο πολλά πράγματα, να ε, δημιουργήσει περισσότερε ερευνητικέ δυνάμει σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί εμεί εδώ μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε, αλλά με τέτοιου είδου συζητήσει δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του και θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένε δράσει. Κανένα δεν μπορεί να αναλάβει δράση εξ ονόματό μα. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε το επόμενο ψήφισμα και το επόμενο ψήφισμα. Ε, όλα αυτά είναι ε, κενά λόγια και δεν θα φτάσουμε τελικά πουθενά. Μία η γυναίκα η οποία έχει υποστεί βιασμό ε, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα σε άμβλωση. Αυτό αποτελεί λύση σε τέτοιου είδου ένοπλε σειράξει, δηλαδή αυτό, αυτή είναι η επιλογή που δίνουμε σε μια τέτοια γυναίκα. Ε, κάθε ε, εμπόλεμη κατάσταση είναι τραγική για μια γυναίκα, αλλά μια άμβλωση σημαίνει βέβαια και ένα παιδί, το οποίο χάνει τη ζωή του και σημαίνει και αντίστοιχη επιβάρυνση για τη γυναίκα. Οπότε δεν μπορεί, εντάξει μπορεί εντό εισαγωγικών να είναι ένα δικαίωμα, αλλά από την άλλη πλευρά η άμβλωση, αλλά από την άλλη πλευρά σίγουρα ε, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι ενδεδειγμένη η βέλτιστη λύση, η άριστη λύση. Κατά τη δική μου άποψη χρειαζόμαστε περισσότερες συνευτικές ε, αποστολές. Θα πρέπει ε, σε αυτό το επίπεδο να αξιοποιήσουμε και τα ε, ε, κονδύλια μας ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση και ακριβώς εδώ θα πρέπει να θέσουμε την, την, την προτεραιότητα, το ειδικό βάρος των δράσεών μας. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ειδικές χώρες και ταυτόχρονα θα πρέπει να αυξήσουμε και την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Ας λοιπόν ε, μεταφέρουμε εκεί που πρέπει ε, την, ε, την έμφαση στο πλαίσιο των συζητήσεων μας. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, μου είπατε να μιλάω λίγο πιο αργά, ζητώ συγγνώμη, απλά με αγγίζει πολύ αυτό το σύνδημα, Ε, αναφέρθηκα λοιπόν στο γεγονό ότι ε, ενδεχομένως να ε, μην ε, επιτυχάνουμε πολλά διοργανώνοντας τη μία ε, μετά την άλλη διάσκεψη γιατί αυτό το, τα, πολύ τραγικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες ειδικότερα ο βιασμός δηλαδή στη σειρά των γυναικών και των κοριτσιών δεν μπορούν να λυθούν με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά τρομακτικό ε, στον 21ο αιώνα να ακούμε ότι λαμβάνουν χώρα ε, μαζικοί βιασμοί. Ε, όλος ο κόσμος γνωρίζει το τι συμβαίνει. Όλοι έχουν ακούσει για τέτοιου είδου μαζικού βιασμού και αν πραγματικά αυτή είναι η διάγνωση, αν γνωρίζουμε ότι πραγματικά όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, τέτοιες φρικαλαιότητες, τότε θα πρέπει ή, ε, να, έχουμε περισσότερες και πιο ενισχυμένες συνευτικές αποστολές από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα ακριβώς στις περιοχές εκείνες όπου λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους βιασμοί και γυναικών. Και αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα εκτάκτως. Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα ε, χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να βοηθήσουμε τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί ένα τόσο τραυματικό ε, ε, ε, δεν χρειάζονται απλώ ανθρωπιστική βοήθεια και τίποτα άλλο. χρειάζονται πιο άμεση βοήθεια. Και δεν συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε από μια συνάδελφο και η οποία ήδη έχει αποχωρήσει από την αίθουσα, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βιασμό να έχουν το δικαίωμα άμεσης άμβλωσης, γιατί μια άμβλωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για, το, ε, για μια τραυματική εμπειρία όπως αυτή του βιασμού. Άλλωστε ας μην ξεχνάω ότι άμπλωση ε, σημαίνει ε, και περισσότερος πόνος για τη γυναίκα και βέβαια θάνατος ενός του παιδιού. Οπότε δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε λύση εδώ η άμπλωση ε, για το βιασμό ή δεν μπορεί να θεωρείται ως τέτοια. Επίσης ε, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν φορείς της, ε, ε, κύριους φορείς της μιας ειρηνευτικής διαδικασίας οι γυναίκες, αλλά αυτό θα λάβει χώρα μόνο εάν πραγματικά γίνει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο δηλαδή πρωτοβουλειών και στι εν λόγω χώρε. Κυρία Μπεσέρα, έχει το λόγο, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί μα πιέζει και ο χρόνο. Να ευχαριστήσω καταρχά τους ομιλητές για την παρουσίασή τους, ε, τα όσα μας είπαν, να μπορούν ε, να ε, εργαστούν με πιο συνεκτικό τρόπο και οι επιτροπές μας και κυρίως η Επιτροπή Γυναικών. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία πράγματα και σας ευχαριστώ κυρία Σούμαχερ που το αναφέρατε αυτό. Το πλαίσιο για αυτή την αναθεώρηση και η χρονική συγκυρία είναι το θεματολόγιο για το 2030 οποιαδήποτε δράση, οποιαδήποτε πρωτοβουλία για μας ε, ε, θα πρέπει να επικεντρώνεται στην, ε, στο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης του 2030. Καταρχάς γιατί υπάρχουν το 5 και το 16 η ισότητα των φύλων, ε, δηλαδή ως ε, ραχοκοκαλιά όλων των δράσεων και κυρίως ο στόχος της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Και σε αυτή την περίπτωση αυτή η αναθεώρηση του 1325 ε, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το νέο ψήφισμα 2242 θα πρέπει να αξιολογούνται για το κατά πόσο είναι κατάλληλα, για το κατά πόσον ε, τηρούνται ε, με βάση το πόσο ε, χρησιμεύουν προκειμένου να τηρήσουμε το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών, όπου είναι ένας από τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Υπάρχουν κάποια αναφυσβήτητα γεγονότα, ότι ο βιασμός, για παράδειγμα, είναι ένα συστηματικό όπλο πολέμου. Έχει σχέση με τον πόλεμο και με τη σύραξη και η σεξουαλική βία έχει άμεση σχέση με αυτό. Πρόκειται για κάτι το οποίο όχι μόνο δημιουργεί μια διάκριση ε, επιφέρει πόνο και μόνιμη ζημία σε κορίτσια και γυναίκες, αλλά επίσης έχει επιπλέον θύματα. Ε, είναι τα παιδιά καρπός αυτών των βιασμών και αφενός είναι σαφές ότι ε, το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες είναι ευάλωτες ε, αυξάνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη και δεν υπάρχουν ε, υπηρεσίες, δράσεις και σεξουαλικής αναπαραγωγής. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε με αυτό το νέο ψήφισμα, οτιδήποτε δεν έχει τηρηθεί με το προηγούμενο ψήφισμα θα πρέπει να τηρηθεί. Ε, παρακαλώ, την ίδια παρατήρηση λίγο πιο αργά να μιλάτε διότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες αυτές, αλλά ίσως ε, αυτό το νέο ψήφισμα επικεντρώνεται πολύ σε πόρους για προστασία και δεν λαμβάνει υπόψη του τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα. Ε, και επίσης όσον αφορά το πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, τήρηση των δεσμεύσεων σε ανθρωπιστικό επίπεδο, ε, για την εγγύηση για μια ασφαλή άμβλωση. Σίγουρα η άμβλωση δεν είναι η λύση, δεν είναι δικαίωμα ε, αυτό καθε αυτό, αλλά η άμβλωση ε, στόχο έχει να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες να προστατευτούν από μια κατάσταση που τους δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Πολλό δε μάλλον άμα προέρχεται από ένα βιασμό το οποίο είναι έγκλημα. Ε, η ανθρωπιστική απάντηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε οι γυναίκες σε περιοχές ε, σύραξης να την χάνουν κατάλληλης προστασίας και, και η πατία πρόσωπος η κυρία Μογκερίνη και ο Επίτροπος Σιλιανίδης μας είπαν ότι πρέπει να εγγυηθούμε αυτό το δικαίωμα. Η γυναίκα ή το νερό κορίτσι το οποίο βιάστηκε και είναι έγκυος λόγω του βιασμού έχει δικαίωμα να λαμβάνει υπηρεσίες και πληροφορίες αναπορυγιογικής ε, υγείας ώστε να μπορεί να αποφασίσει και να έχει τη στήριξη που πρέπει ε, ώστε να μην συνεχίσει να υποφέρει. Δεν σημαίνει αυτό οπωσδήποτε άμβλωση, ούτε είναι υποχρεωτική η άμβλωση, ούτε θα υποχρεωθούν ε, να ε, προχωρήσουν σε άμβλωση, αλλά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να επιλέξουν τι είναι αυτό το οποίο θα μειώσει τον πόνο τους. Και επίσης ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ στην Επιτροπή μας, ε, την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο για να προστατέσουμε τις γυναίκες σε περιοχές πλησίρεξης. Μπορείτε να ολοκληρώσετε και ολοκληρώνω με αυτό. Ολοκληρώνω λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε να ζητούμε την υπογραφή και την κύρωση της συνθήκης της ε, Κωνσταντινούπολη για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν την έχουν ακόμα κυρώσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει και να υπογράψει αυτή τη σύμβαση που θα πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό της. Ευχαριστώ. Ε, φοβάμαι ότι ο χρόνο που είχαμε διαθέσει για τη συνεδρίασή μα έχει ήδη περάσει και θα ήθελα να ολοκληρώσω. Ε, δύο φράσεις να πω. Δεκαπέντε χρόνια από την έγκριση του ψηφίσματος 1325 των μέλλον Εθνών. Έκτοτε έχουμε ε, νομοθετήσει επανειλημμένος. Θα ήθελα εδώ να χρησιμοποιήσω ω παράδειγμα τον βιασμό των γυναικών και των κοριτσιών. Πλέον αναγνωρίζεται ω έγκλημα πολέμου. Και αν συμφωνήσουμε ότι οι ένοπλε σειράξει. και νομίζω ότι από αυτού συμφωνούμε ότι η ένοπλη σύραξη είναι το υπέρτατο κακό για οποιαδήποτε οικογένεια, για οποιαδήποτε γυναίκα, για οποιοδήποτε παιδί, για οποιοδήποτε ηλικιωμένο, για όλου και κατόπιν Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να συλληφθούν οι δράστες και να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να σταματήσει αυτό το έγκλημα πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Δεν θα πρέπει να αφιστούμε προσπαθειών. Κύριε Καμιλέρη, έχετε εξαιρετική πείρα με την αποστολή Αταλάντα. Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης ήταν ακριβώς ότι συνελήφθησαν οι πειρατές και μπορέσαμε να τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό αποτελεί ε, στοιχείο αποτροπής κατά της πειραπητίας στο κέρας της Αφρικής. Και θα πρέπει να μιλήσουμε και για μέτρα προκειμένου να σταματήσει η ατιμορρησία με το να ε, προσάγονται ενώπιον των δικαστηρίων οι δράστες. Πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, προσπάθειές μας για την ειρηνευτική διαδικασία. Συμφωνώ δε με την κυρία Βισνέσκα Θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ε, το να επικεντρωθούμε συγγνώμη, στο δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι λύση. Απλώς ε, θα έρθει να προσθεθεί στον πόρνο των θυμάτων. Το πρόβλημα είναι να ε, αποτελεσματικά ειρηνευτικές αποστολές ε, και δυστυχώς εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών υπήρχαν ε, ήδη κάποια πολύ άσχημα παραδείγματα να μην αναφερθώ στην ε, δημοκρατία στη, συγγνώμη, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία και τα περιστατικά σεξουαλικής βίας θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και εδώ ε, είναι πρόσδεκτες οι προστάσεις σας κύριε Καμιλέρη ώστε να ε, γίνουν σωστά όλα θα πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτό ολοκληρώνεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ.